guten Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή χρονιά σε όλους. Σας εύχομαι, επαναλαμβάνω και στα γερμανικά ο πρόεδρος, σας εύχομαι καλή χρονιά αγαπητοί συνάδελφοι. Μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, εκπρόσωποι της Κομισιόν, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Ελεκτού Προϋπολογισμού για το 2014. Σας ευχόμαστε και προσωπικά κάθε υγεία και ευτυχία και επίσης και χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική υγεία στα ευρωπαϊκά θεσμικά ιδρύματα. Έχουμε τώρα μια προσθήκη στην ημερησία διάταξη. Είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε μια γρομοδότηση ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων για την Τρόικα. Δυστυχώς δεν υπήρξε η δυνατότητα αυτό να το μάθουμε, να το συμφωνήσουμε γέρος με τη γραμματεία της Επιτροπής ΕΚΟΝ και επομένως Ε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Γραμματεία για να μπορέσει να προετοιμαστεί αυτό το έγγραφο εργασίας για γνωμοδότηση μέσα σε τρομερά γρήγορο χρονικό διάστημα. <clears throat> Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό στη συνάντηση των συντονιστών. Και θα σας υπενθυμίσω ότι θα είναι σχετικά σύντομη αυτή η συνάντηση γιατί σας προσκαλώ και σε ένα μικρό κοκτέιλ, σε μια μικρή δεξίωση επί τη ευκαιρία του νέου έτους. Ένα έτος βέβαια το οποίο θα απαιτήσει από μας εντατική εργασία και γι' αυτό αυτή η μικρή δεξίωση η οποία θα λάβει χώρα στις 12.30 μετά από την όπως σας είπα ελπίζω σύντομη συνάντηση των συντονιστών <clears throat> ελπίζω ότι θα είναι θα είσαστε παρόντες σε αυτή τη σύντομη δεξίωση. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη ημερήσια διάταξη, αν συμφωνείτε, για την προσθήκη αυτής της ε, έκθεσης για την Τρόικα. Ε, μπορούμε να την συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη. Μεταδίδεται η συνεδρίασή μας και στο διαδίκτυο και μπορούμε να ξεκινήσουμε στο πρώτο θέμα που είναι η διαδικασία απαλλαγής. Σημείο 3 είναι η απαλλαγή για το 2012 για την ε, Ευρωπαϊκή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είμαστε εμείς η αρμόδια επιτροπή επί της για το θέμα αυτό και έχω την ευκαιρία να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάρτον, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια των Ενεργειών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας κυρία Μπάρτον και επίσης από το ε, ελεκτικό συνέδριο είναι ο κύριος ε, Στόκ παρόν. Μποστόκ, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε. <clears throat> Η συγητής είναι ο Γιάνν Μίλντορ. Θα ήθελε ο εισηγητής να λάβει το λόγο τώρα ή αργότερα. <clears throat> Μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο. Και δίνω το λόγο στον ε, κύριο Μποστόκ. Είναι κάποιος ε, παρόν από το <clears throat> ελεκτικό συνέδριο που θα λάβει το λόγο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου. Τότε ίσως <clears throat> προτείνω να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στην κυρία Μπάρτον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προβλέπεται βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας με αρμοδιότητες οι οποίε έχουν σαν αποτέλεσμα να παίρνουμε την πολιτική μας δουλειά πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν και συμμετέχουμε και εμείς στη διαδικασία απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη, αν και δεν είναι κάτι που απαιτείται απόλυτα από εμά. Και υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να σας ε, αναφέρω πράγματα σχετικά με αυτά που έχετε αναφέρει και εσείς παλιότερα στην Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα όμως σας κοιτάξουμε λίγο πριν από το 2012, τη χρονιά δηλαδή για την οποία είναι η απαλλαγή, γιατί η χρονιά αυτή, το 2012 δηλαδή, είναι μια μεγάλη επέτειος. Είναι 50 χρόνια από τότε που άρχισε να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις χώρες ε, Ειρηνικού, Αφρικής και Καραϊβικής. Πάνω από 1.300 σχέδια σε 92 χώρες λοιπόν έχουμε χρηματοδοτήσει 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή συνολικά. 53 εκατομμύρια ήταν τεχνική αρρωγή. 4 δισεκατομμύρια για ενεργειακά προγράμματα και 1,4 για το είδωρ και την υγεία. Από το 2003 η τράπεζά μας ε, λειτουργεί στην περιοχή αυτή βάσει της εταιρικής σχέσης Κοτονού για τα υπερπόντια διαμερίσματα. Η χρηματοδότηση στις χώρες ΑΚΕ έρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ σήμερα. Όμως πέρα από τους ίδιους πόρους της τράπεζας που δανειζόμαστε εμείς από τις κεφαλαιαγορές με εγγύηση από τα κράτη-μέλη, Βάσει της Κοτονού η νέα εξέλιξη ήταν ότι οι χώρες ΑΚΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα βάση της επενδυτικής διευκόλυνσης της Κοτονού. Είναι ένα ταμείο 20 ετές με 3,2 δισεκατομμύρια. Η χρηματοδότηση λοιπόν των επενδυτικών αναγκών γίνεται βάσει μέσων ευελιξίας και αποτελεί καταλήτη για να προσελκυθούν και άλλοι επενδυτές, μακροπρόθεσμα και ντόπιοι. Είναι, συμπληρώνονται όλα αυτά και με χρήματα από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε τα προγράμματα να λάβουν πραγματικά χώρα ή τέλος πάντων προκειμένου να ενισχυθεί η αξία τους. Το 2012 παγιώσαμε ακόμα περισσότερο τη στρατηγική μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας και ε, ενισχύσαμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μικρών επιχειρήσεων ε, κυρίως σε τομείς όπως είναι το κλίμα, η ενέργεια. Συνεχίσαμε να επικεντρωνόμαστε στο δημοσιονομικό τομέα με πιστώσεις θα επανέλθω σε αυτές και βάσει των εξελίξεων στο τραπεζικό τομέα δώσαμε μεγαλύτερη σημασία ακόμα στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές πάνω στο κλίμα και το περιβάλλον. Το 2012 ο συνολικός δανεισμός ήταν 644 εκατομμύρια. 41 εκατομμύρια τεχνικής αρρωγής 21 προγράμματα σε 9 χώρες, σε 4 ομάδες χωρών. Και ένας τομέας με τον οποίο έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν είναι πώς συνεργαζόμαστε με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 50 ε, χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματά μας. 119 προγράμματα δηλαδή τελικά συγχρηματοδοτήθηκαν. Το 1 τέταρτο, και αυτό είναι και ο στόχος μας των προγραμμάτων δηλαδή, είχαν ε, στοιχεία σχετικά με το κλίμα και είναι το 22% του συνολικού δανεισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη στις υπανάπτυξη χώρες. Η τράπεζα λοιπόν αύξησε το δανεισμό της βάσει της δανειστικής διευκόλυνσης αναλαμβάνοντας περισσότερους κινδύνους. Ο όγκος διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά από 193 δισεκατομμύρια στα 255 το 2012. Έτσι φτάσαμε σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια συνολικά. Κάτι το οποίο διασφαλίζει ότι οι πόροι τελικά έχουν πολλαπλασιακό αποτέλεσμα και χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς. Θέλω εδώ να αναφερθώ σε κάποια προγράμματα για να σας εξηγήσω πιο συγκεκριμένα που πάνε αυτά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον οποίο και μας ρωτάτε. Το παράδειγμα των μικροπιστώσεων. Οι χώρες της Ανατολικής Αφρικής επωφελούνται κυρίως προκειμένου να στηρίξουν την ε, αντίστοιχη αγορά τους και για αυτά τα προγράμματα θα σας δείξω τώρα ένα μικρό βίντεο, στο τέλος μάλλον, για να σας δώσω να καταλάβετε ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Κάπου 90.000 θέσεις απασχόλησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εποφελήθηκαν. Ένα άλλο πρόγραμμα, εκείνο της ιδιωτικής διευκόλυνσης στην Κένια χρηματοδοτεί την επέκταση και τον εξυγχρονισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Κάτι που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα εκεί. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά μεσοπρόθεσμα το ωφέλη θα είναι μεγαλύτερα. 50.000 θέσεις απασχόλησης περίπου θα δημιουργηθούν σε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το τρίτο πρόγραμμα, μια καινοτομία, κάτι που ζητήθηκε κατά το παρελθόν, είναι ότι ο κόσμος ζητάει να χρησιμοποιούνται περισσότερο εγγύησεις για την υποστήριξη προγραμμάτων. Δουλεύουμε το FC για πρώτη φορά και έχουμε μια νέα διευκόλυνση εγγύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρει τη στήριξή μας σε τράπεζες που θέλουν να βοηθήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε πολλές τράπεζες στην Αφρική δεν θέλουν να αναλάβουν τον κίνδυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε εμείς τις στηρίζουμε. 25.000 θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν έτσι. Υποδομές. Η τράπεζα έδωσε 360 εκατομμύρια για 9 μεγάλα προγράμματα υποδομών. 250 εκατομμύρια για προγράμματα παντού στην Αφρική. 750 ΜΒ παραπάνω στο, στη δύναμη του ηλεκτρισμού εκεί. Στην Αιθιοπία για παράδειγμα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Με τα προγράμματα αυτά 400.000 κατοικίες ή επιχειρήσεις στην Ήπεθρο είτε θα συνδεθούν και θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για πρώτη φορά ή θα επωφεληθούν από πιο καθαρή ενέργεια από ό,τι είχαν κατά το παρελθόν. Κάτι το οποίο δίνει νέες οικονομικές ευκαιρίες. Στο Καμερούν, επίσης, προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης έχουν σαν αποτέλεσμα να αλλάξει και εκεί η κατάσταση όσον αφορά τις ηλεκτρικές πηγές τους και φυσικό αερίου. Και αντιμετωπίζεται το θέμα της μεταβλητότητας της εποχιακής. Επίσης, ένα φράγμα ε, στο ποταμό Σανάγκα. Θα αυξήσει την παραγωγικότητα των ε, εργοστασίων ε, εκεί ηλεκτρισμού και θα υπάρξει σύνδεση για 2.400 παραπάνω περιοχές στην Ήπεθρο. Επίσης, θα υπάρξουν και άλλα προγράμματα για παραγωγή ενέργειας. Έτσι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης και έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Τώρα στις χώρες όπου έχει υπάρξει σύγκρουση, εκεί βέβαια είναι πιο δύσκολο για μας να επενδύσουμε εξαιτία του κινδύνου. Ε, ακτή ελεφαντοστού, Κινέα, εκεί χρηματοδοτούμε πάλι προγράμματα ηλεκτρισμού που οδηγούν σε σύνδεση με το μεγάλο εργοστάσιο στη Δυτική Αφρική πολύ βασικό για την περιοχή και μειώνεται και το κόστος της ενέργειας. Πολύ σημαντικό για πολλές φτωχές χώρες, γιατί χωρίς ενέργεια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επιπλέον από το δάνειο των 95 εκατομμυρίων υπάρχει και τεχνική αρρωγή για την Δυτική Αφρική και από την τραπέζα μας και από το Trust Fund της περιοχής εκεί που συμπληρώνεται και με συγχρωματοδότηση από άλλες πηγές. Το 2012 η τράπεζά μας έδωσε 160 εκατομμύρια σε πέντε προγράμματα σχετικά με το κλίμα στον ενεργειακό τομέα τέσσερα μεγάλα προγράμματα για να αντικατασταθούν τα ορυκτά από άλλα υλικά για την παραγωγή ενέργειας. Μεταξύ άλλων Γαλλική Πολυνησία. 7,5 εκατομμύρια ήταν το δάνειο από την τράπεζά μας για ένα μεγάλο εργοστάσιο εκεί για να μειωθεί εκεί το κόστος της ενέργειας και για να εγκατασταθεί σύστημα air conditioning κλιματισμού. Θέλω επίσης να αναφερθώ λιγάκι και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε περιοχές που έχουμε αναφέρει και παλιότερα. Σε αυτά που σας είπα μέχρι τώρα φαίνεται ότι σας δίνω λεπτομέρειες για το τι αποτελέσματα μπορεί κανείς να περιμένει από τη δράση της τράπεζας. Και γιατί, γιατί το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά όπου αρχίσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης αποτελεσμάτων μέτρησης αποτελεσμάτων, προκειμένου να έχουμε δηλαδή μια μεθοδολογία με πραγματικά ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η πρώτη τέτοια έκθεση δημοσιεύθηκε και φαντάζομαι ότι μπορείτε και εσείς να έχετε ένα αντίγραφο και εκεί φαίνεται η ανάλυση των δράσεων που αναλάβαμε και που βελτιώσαμε την κατάσταση αυτή τη χρονιά. Με δύο λόγια, οι οχτώ περιπτώσεις που μελετήσαμε. Τι δείχνουν. Δείχνουν Πρώτα απ' όλα και φέτος θα επαναληφθεί το ίδιο, αλλά τι δείχνουν όλα αυτά. Ότι ήδη υπάρξει ε, μεγαλύτερη και καλύτερη επιλεξιμότητα των προγραμμάτων ώστε το όφελος να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο. Και αυτό αντιστοιχεί στην εντολή η οποία έχει συμφωνηθεί με όλους τους συμμετέχοντες. Εννοείται ότι μαθαίνουμε πολλά μαθήματα από την πιλωτική φάση του 2012 και σίγουρα θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη μεθοδολογία μέτρησης αποτελεσμάτων. Και τα μαθήματα που μαθαίνουμε τα μεταφέρουμε στην ομάδα εργασίας βέβαια. Όσον αφορά τη διαφάνεια τώρα, και εδώ είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, η διαφάνεια είναι ένας τομέας για τον οποίο συχνά μεστάται να κάνουμε περισσότερα. Εδώ λοιπόν έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα το φθινόπωρο όταν συμμετείχαμε και εμείς στην ε, πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την γραμματεία της οργάνωσης αυτής για τις προδιαγραφές. Την προηγούμενη φορά είχα πει ότι οι προδιαγραφές δημιουργούνται όσον αφορά τα δάνεια που δίνουμε, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προδιαγραφές και για άλλες περιπτώσεις. Συνεπώς, στην επόμενη φορά που θα συναντηθεί η ομάδα αυτή εργασίας θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις προδιαγραφές. Όσον αφορά τώρα την πολιτική μας ε, κατά της ε, διαφθοράς. Συνεχίζουμε με την προσέγγισή μας που είναι μηδέν ανεκτικότητα, με νέα όμως εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Η πολιτική για την καταγγελία, ε, όσον αφορά την ε, μελέτη ακεραιότητας, άλλες διαδικασίες που εφαρμόζουμε. Και βέβαια χρησιμοποιούμε και μια νέα γλώσσα όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Προχωρήσαμε περισσότερο και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης υπέρ των πελατών μας τους δίνουμε χρηματοδότηση για πιο μακροχρόνια προγράμματα βασιζόμενες στις νέες διαδικασίες. Έχουμε 30 προγράμματα σήμερα σε συνεργασία και μπαίνουμε και σε νέες περιοχές της Ασίας και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, πέρα δηλαδή από τις χώρες ΑΚΕ. Έχουμε συνεργαστεί περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν και σε θέματα προγραμματισμού με άλλους. Τώρα μπαίνουμε στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε και με την Κομισιόν και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργαζόμαστε για τον προγραμματισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ, για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ένα τον άλλον πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα. Ένας από τους τομείς κλειδί για τον οποίο μας έχετε ερωτήσει κατά το παρελθόν, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συνέργεια, είναι οι εξωτερικές υπηρεσίες της τράπεζάς μας, πώς συνεργάζονται με τις αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει χρόνο για να αποδώσει. Πάντως, και εδώ προχωράμε. Έχουμε ήδη τέσσερα γραφεία στο Πεκίνο, στο Κίεβο, τη Μόσχα και το Σάντο Ντομίνγκο, όπου είμαστε στο ίδιο κτίριο με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπάρχουν και άλλες 7 χώρες όπου θα χρηματοδοτήσουμε μια τοπική υπηρεσία. Μέχρι τώρα η παρουσία μας είναι πολύ περιορισμένη στον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα δράσεων ε, που, όπου ελοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά από την άλλη μεριά τα αποτελέσματα ανάπτυξης θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Πρόκειται για 400 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο 2013 βάσει του 10 ου Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Ένα από τα πολύ σημαντικά προγράμματα για τα οποία σίγουρα θα σας μιλήσουμε πολύ στο μέλλον. Οι υποδομές ε, λοιπόν και ο χρηματοδοτικός ταμέας είναι από τους βασικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμεθα. Αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε όμως με αυτό το τελευταίο είναι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις χώρες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Κατά το παρελθόν ήταν δύσκολο για μας να δουλέψουμε στις πιο φτωχές χώρες, εκείνες που πλήττονται περισσότερο από συγκρούσεις, ε, χώρες ασταθείς, ε, κλπ. Εδώ τώρα περιμένουμε ότι θα αυξηθεί η δανειστική μας δραστηριότητα και σε τέτοιες περιοχές χρησιμοποιώντας νέα καινοτόμα μέσα εγγύσεων. Και η τράπεζά μας θα ψάξει να βρει ευκαιρίες ακόμα περισσότερο με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει βέβαια του προπολογισμού που διαθέτουμε. Θα ολοκληρώσω τονίζοντας ότι η τράπεζά μας στοχεύει η επενδυτική διευκόλυνση να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία και με τις χώρες ΑΚΕ και με νέους εταίρους. Και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα δείτε τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Φέτος η καινοτομία είναι... Ξέρω ότι συχνά ρωτάτε πολλές φορές τι κάνουμε με τα προγράμματά μας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, λοιπόν, αυτή τη φορά σας φέραμε ένα πολύ σύντομο βίντεο για να σας δείξουμε τι κάνουμε με τα προγράμματα ε, μακροπιστώσεων, μικροπιστώσεων μάλλον, στην ε, Δυτική Αφρική. Φτάνει λοιπόν να πατήσουμε το κουμπί για να δείτε το βίντεο αυτό. Στο μέλλον ίσως να μπορέσουμε να έχουμε και επικοινωνία με Skype, κάποιο τρόπο τέλο πάντων ανάμεσα σε εσά και του όσους έχουν υποφεληθεί από τέτοιες μικροπιστώσεις. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε μια άλλη φορά να μπορέσετε να δείτε τα προγράμματά μας από πιο κοντά. Πάντως προς το παρόν σήμερα μόνο αυτό, το μικρό βίντεο που σας έφερε. Ευχαριστώ.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 Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Κυρία Μπάρτον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκθεσή σας. Το ελεκτικό συνέδριο δυστυχώς δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σήμερα, γιατί έχουμε μια σημαντική εσωτερική συνάντηση σήμερα. σε ό,τι αφορά την επιλογή, την εκλογή ενός νέου Προέδρου για το ελεκτικό συνέδριο. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό και πρέπει να αποδεχτούμε την απουσία τους, οπότε στρέφουμε προς τα μέλη της Επιτροπής μας. Και φυσικά ο κύριος Μίλτορος, εισηγητής, έχει πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είδα το βίντεο με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ πέντε χρόνια έχω ζήσει στην Κένια Ε, δεν θα σας μιλήσω βέβαια στην ε, γλώσσα τους, ε, παρά το γεγονός ότι μπαίνω στον πειρασμό. Ήταν πολύ ενημερωτικό αυτό το βίντεο. Κάτι πρέπει να γίνει με το εμπόριο πολύτιμων λίθων στο Ναϊρόμπι. Ε, που είναι ένα από τα βασικά θέματα. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως είδαμε και από το ε, βίντεο, έχουν μια πολύ καλή ενημερωτική πολιτική και από ό,τι είδα και από τα έγγραφα τα οποία έλαβα, είναι δύσκολο να βρεθούν σφάλματα. Από ό,τι βλέπω είναι μια ιστορία επιτυχίας Τουλάχιστον αυτό κρίνω βάσει των πληροφοριών που έλαβα. Δεν σημαίνει ότι τίποτε δεν πάει ποτέ στραβά. Η Νιγηρία, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ε, περίπτωση. Δεν λέω βέβαια ότι αυτό είναι ανακουφιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να απομονώσω από τις υπόλοιπες ιστορίες επιτυχίας. Τα υπόλοιπα ζητήματα παραμένουν. Πρώτον, Ε, εκεί PMG ε, είναι ε, ο εσωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ίσως θα έπρεπε να τους ακούσουμε και εκείνους κάποια στιγμή. Μία γενικότερη ερώτηση, γιατί όπως σας είπα έχω ζήσει στην Αφρική ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλά προγράμματα, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ε, υλοποιεί προγράμματα, υπάρχουν και πολλοί άλλοι οργανισμοί που υλοποιούν προγράμματα εκεί. Κάποια βέβαια δεν προχωρούν τελικά και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς γίνεται η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, ε, με την Τράπεζα ε, ε, Ανάπτυξης της Ασίας, πώς γίνεται η συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς. Το θέμα των μικροπιστώσεων αυτή τη στιγμή είναι αρκετά επίμαχο. Οι ιστορίες που ακούει κανείς για τις μικροπιστώσεις πραγματικά ανοίγουν την όρεξη. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της ε, ΕΤΕΠ. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ακούσει ότι αυτές οι συνεργασίες αποτυγχάνουν και τα προγράμματα αποτυγχάνουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, για παράδειγμα στην περίπτωση της Νιγηρίας υπάρχει υποψία απατών, αλλά πέρα από αυτό μπορεί απλώς να αποτύχει ένα πρόγραμμα. Για, τα, για το ε, Ταμείο Επενδύσεων ε, στην Αφρική. Ποιο είναι το επίπεδο, ποιο είναι το ποσοστό ε, εφαρμογής. Υπάρχει αύξηση, πώς είναι η κατάσταση σε σχέση με το ποσοστό αυτό. Και επίσης η χρήση των ε, ιδίων πόρων ε, στην Αφρική. Για παράδειγμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης δραστηριοποιείται κυρίως στην Αφρική. Οπότε υπάρχει καμία διαφορά ως προς τα αποτελέσματα αν ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει παρουσία διεθνών οργανισμών, ποια γίνεται η πώς γίνεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι διαφορετικές οι δικές μας προδιαγραφές από των άλλων τραπεζών, ποιες είναι οι βασικές διαφορές που ε, διαπιστώνεται και... Πιστεύετε ότι οι προδιαγραφές της Ένωσης είναι καλύτερες από των υπολείπων, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να τις υπερασπιστούμε. 3,363 εκατομμύρια είναι η δανειοδότηση στις χώρες ΑΚΕ τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε ε, θα ήθελα να μου πείτε πόσα από αυτά ήταν ανακτήσιμα, ε, πώς έχει εξελιχθεί ε, το Ταμείο κατά τη διάρκεια των ετών. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επίσης, ε, δεν καλύφθηκε το Ταμείο Επενδύσεων από, την ε, Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υποστήριξης των Ιδιωτικών Προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των 2013. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα σήμερα, αλλά επειδή είναι ε, σημαντικό το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ε, θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε. Η ανάμιξη. Επειδή υπάρχουν πολλά εργαλεία, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί συνήθως ε, υπάρχει μια αρχή που αναλαμβάνει τα προγράμματα και πώς γίνεται ο έλεγχος της αρχής αυτής γιατί δεν υπάρχει μόνο ε, δεν υπάρχει το κονδύλια μόνο της ΕΤΕΠ, υπάρχουν και άλλα κονδύλια που εισραίουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται λοιπόν ε, η συνεργασία, ο έλεγχος, ε, υπάρχουν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί που έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου. Τα δικά τους εργαλεία είναι καλύτερα από τα δικά σας. Και μπορεί να σας λένε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται να μας κάνετε πολλές ερωτήσεις, πρέπει απλώς να μας πιστέψετε. Βλέπω ότι ως προς το Ταμείο Επενδύσεων, από ό,τι βλέπω, έχετε ε, ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους ε, ύψους μισού δισεκατομμυρίου. Αυτό είναι μια κανονική κατάσταση, είναι κάτι το εξαιρετικό, πώς το χαρακτηρίζετε. για την, ε, το πλαίσιο μετρήσεων των αποτελεσμάτων, ε, το, ε, Πώς, πότε μπορείτε να το κάνετε, η αξιολόγηση πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει την πρώτη χρονιά, σε ποια φάση θα είστε σε θέση να μας δώσετε μία, να μας κάνετε μία δήλωση ότι είναι ένα πραγματικά τέλειο σύστημα. Νομίζω ότι έτσι ολοκλήρωσα τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο συνάδελφο που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο καταρχήν της Κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Είναι ο Διευθυντής ο κύριος Ρομπέρτο Ριτόλβι και ο Χάιμις Φρέις Κόντε. Ποιο θα λάβει το λόγο από του δύο σα Ο επικεφαλής ε, μονάδο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο πρέπει να σας πω είναι ότι η διευκόλυνση επενδύσεων για τις χώρες ΑΚΕ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την Κομισιόν για την υποστήριξη των ιδιωτικών τομέα στις χώρες αυτές. Με ικανοποίηση βλέπει η Κομισιόν τις προόδους οι οποίες επετέθησαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά το πλαίσιο καταμέτρησης αποτελεσμάτων και συνεχίζουμε την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ο κατάλληλος αντίκτυπος για τις χρηματοδοτήσεις αυτές που δίνονται στις χώρες ΑΚΕ. Η Κομισιόν προσπαθεί να συμμετέχει με ενεργό τρόπο στις αξιολογήσει των σχεδίων που ε, υποβάλλονται από τη διευκόλυνση επενδύσεων της ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και να τη συμπληρώνει με χρηματοδοτικές δράσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η Κομισιόν επίσης είναι παρούσα και διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε κάθε πρωτοβουλία επενδύσεων και αυτό ήταν μια βασική σύσταση που είχε διατυπωθεί το 2010 και η Κομισιόν εξάλλου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου βέβαια στη διαδικασία αποφάσεων για την επενδυτική αυτή διευκόλυνση για τις χώρες ΑΚΕ. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία <clears throat> του πλαισίου για την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων γιατί για τις δραστηριότητες του λεγόμενου blending της ε, ε, ανάπτυξης κοινών δράσεων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναπτύξει αυτό το σύστημα καταμέτρησης για τα αποτελέσματα και έχουν δημιουργηθεί κανόνες, διαδικασίες και αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζονται και από άλλα χρηματοδοτικά όργανα στα πλαίσια δράσεων που χρηματοδοτούν από την Κομισιόν στα πλαίσια αυτής της ενέργειας του blending. Είναι λοιπόν σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία και εξάλλου νομίζω ότι μπορούμε να επωφεληθούμε από τις προόδους οι οποίες έχουν επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για να μπορέσουμε και εμείς να διαμορφώσουμε ένα γενικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να έχουμε ένα πλήρες και ε, γενικό όραμα σε ό,τι αφορά τις δράσεις της Κομισιόν στο blending με τα άλλα χρηματοδοτικά όργανα. Προτού κλείσω θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό που έθεσε ο κ. Μούλτερ και να τονίσω και πάλι ότι έχετε δίκιο. Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος για το θέμα αυτό αυτής της έκθεσης. Αν η έκθεση Κομισιόν για το ιδιωτικό τομέα δεν αναφέρεται στο επενδυτικό αυτό εργαλείο, στη διευκόλυνση για επενδύσεις της χώρας ΑΚΕ, αυτό είναι σαφές ότι πρέπει να διορθωθεί. Και στην επόμενη έκθεσή μας θα πρέπει <clears throat> να αναφέρεται αυτή η μνήα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μπάρτον να απαντήσει αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ <clears throat> για να απαντήσω. Αν υπάρξει κάτι το οποίο θα μου ξεφύγει, είμαι στη διάθεσή σας για να επανέλθω. Για τα μποτιλιαρίσματα στην Αϊρόμπη θα πρέπει να επανέλθουμε. Έχουμε χρηματοδοτήσει τον υπόγειο σιδηρόδρομο σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές. Προσπαθούμε να έχουμε μια βιώσιμη δυνατότητα δημοσίων συγκοινωνιών στην Αϊρόμπη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι να πούμε ότι όλα πάνε καλά, όπως είπατε αλλά μερικές φορές δημιουργείται εντύπωση ότι όλα πάνε στραβά. Και θέλουμε για αυτό το λόγο να εξηγήσουμε ότι τα περισσότερα από τα χρήματα τα οποία εσείς θέλετε να ελέγξετε πιάνουν τόπο. Φυσικά στις αναπτυσσόμενες χώρες <clears throat> τα πράγματα παίρνουν πολλές μορφές. Όταν βρισκόμαστε στην αρχή των δημοσιονομικών προοπτικών, βλέπετε να υπάρχει μεν ενδιαφέρον στην Αφρική, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη κλίμακα επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί υπάρχει διστακτικότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο και στον τοπικό ιδιωτικό τομέα. Πολλές φορές υπάρχει μια λανθασμένη αντιμετώπιση από τους ιδιωτικούς επενδυτές για τη σημασία και τα σχέδια που αναπτύσσονται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επενδυτικό αυτό εργαλείο τη διευκόνηση, εφόσον θέλουμε να είναι ανανεούμενα τα κονδύλια, θέλουμε <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και επαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσει να γίνει πιο βιώσιμη αυτή η ενέργεια. Μόνο 3 ή 4% είναι το ποσοστό αποτυχίας των σχεδίων μας. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Και γι' αυτό Ε, επειδή ακολουθήσαμε ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο περιορίζει τον κίνδυνο, θεωρούμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει μπορούμε, αν έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να έχουμε και μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, μια κερδοφορία 5% και σε ό,τι αφορά τον, ε, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα θα μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε τρεις φορές αυτά τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2020 και μετά θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα ακολουθήσει αν θέλουμε μια πιο μεγάλη κλίμακα επενδύσεων. Για το λογιστικό έλεγχο από την KPMG και άλλες εταιρείες, <clears throat> ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στην ιστοσελίδα μας και λυπάμαι βέβαια που δεν είναι παρόν το ελεκτικό συνέδριο, γιατί με την τριμερή συμφωνία είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των σχεδίων μας και έχουν δει την ε, διαχείρισή μας για το καταπίστευμα για την ανάπτυξη υποδομών στην Αφρική, για τις χώρες ΑΚΕ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψή τους για τα θέματα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία μεταξύ σας, το Ελεκτικό Συνέδριο έχει πρόσβαση σε όλα τα σχέδιά μας. Αυτό είναι μια συμβατική μας υποχρέωση σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορούν να πάνε οπουδήποτε και να ελέγξουν οτιδήποτε θέλουν και κάποιοι ιδιωτικοί επενδυτέ δεν δεχτήκαν χρηματοδότηση γιατί δεν θέλαν τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Ρωτήσατε για το ποσοστό απόρριψη. <clears throat> Υπάρχουν πολλοί λόγοι και σε αυτήν την περιοχή και αλλού που κάνουν ένα ελπιδοφόρο σχέδιο να μην μπορεί να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν μονάχα χρηματοδοτικά θέματα, αλλά υπάρχουν και θέματα βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν πολλές φορές σε απόρριψη σχεδίων. Λέτε ότι υπάρχει μεγάλος συνοστισμός για την έγκριση προγραμμάτων και σχεδίων. Υπάρχουν πολλά σχέδια τα οποία χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο που εμείς μπορούμε να υπομισθούμε τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι γίνεται συνοστισμός. Υπάρχουν πολλά σχέδια τα οποία έχουν ε, κάποιες προοπτικές, αλλά για λόγους ε, δημοσιονομικούς πρέπει να τα απορρίψουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τομείς όπου τα πρότυπά μας είναι πιο αυστηρά. Και αυτό επηρεάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ε, σχεδίων. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει υπόψη την περιβαλλοντική πτυγή, ιδίως στις δράσεις εναντί της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να λαμβάνω αυτά πάντα υπόψη σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σχέδια γιατί υπάρχουν οι επιρρογνώμονες οι οποίοι κρίνουν κατά πόσο από πλευρά κλιματικής, αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής τα σχέδια αυτά είναι πρόσφορα. Ένα άλλο θέμα είναι οι δημόσιες προμήθειες και εδώ οι κανόνες θεσπίζονται από την Κομισιόν και βλέπουμε πολλές φορές ότι άλλα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να χρηματοδοτήσουν εκεί που εμείς δεν μπορούμε να το πράξουμε. Εγώ βλέπω μερικές φορές ότι τα, τα πρότυπα μας για προμήθειες είναι αναντίστοιχα με τις ανάγκες αυτών των περιοχών, μπορεί να ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ίσως όχι δεν είναι πρόσφορα για αυτές τις περιοχές και άλλες περιπτώσεις είναι συγχρηματοδότηση με τοπικούς ομίλους και επιχειρήσεις που για λόγους φορολογικούς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όταν υπάρχει κίνδυνος για έκπληση χρημάτων κτλ. Και το θέμα βέβαια της προσθέμενης αξίας είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ διαφέρουμε ιδιαίτερα με τους άλλους διεθνείς χρηματοδότες για το θέμα αυτό. Απλώς οι άλλοι χρηματοδότες μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και να είναι έτοιμοι να υπομισθούν περισσότερο κίνδυνο από ότι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι η Κομισιόν απήντησε στο ερώτημά σας για την έκθεση. Λέτε πώς Ρωτάτε τώρα πώς διατηρείται η ταυτότητα της τράπεζάς μας μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου blending. Βέβαια αυτή η πλατφόρμα του blending της ε, ανάμειξης κονδυλίων έχει σημασία και εν του μέλλοντος. Αλλά όταν υπάρχουν πολλοί χρηματοδότες υπάρχει πάντα ένας επικεφαλής ο οποίος αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη. Και όλα αυτά γίνονται με τον έλεγχο του δημοσιονομικού κανονισμού και η Κομισιόν εξασφαλίζει ότι θα ελέγχονται πλήρως. Νομίζω λοιπόν από αυτή την άποψη το θέμα του ελέγχου είναι επαρκώς αντιμετωπισμένο. Επίσης για τις ταμιακές ροές ποικίλουν από μία χρονιά στην άλλη και είπατε ότι δεν ξέρετε πότε θα αποφέρουν καρπούς όλα αυτά τα σχέδια και πότε θα δείτε ότι πράγματι έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα. Αυτό εξαρτάται και από τη διάρκεια των σχέδιων. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το τελικό τους και το ουσιαστικό τους αποτέλεσμα παρά μόνο μετά από το πέρας των σχέδιων αυτών. Και γι' αυτό έχουμε πόρους για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται μετά από τα σχέδια αυτά. ίσως τα πρώτα σχέδια που θα μπορέσετε να δείτε την ε, περάτωσή τους θα είναι σε 2-3 χρόνια και μετά θα χρειάζεστε άλλα 2-3 χρόνια για να δείτε τους, ε, τα πραγματικά ωφέλη τα οποία προήλθαν από αυτά. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Μπορείτε να δείτε όμως ήδη τι α, ε, θα προκύψει από τις εκτιμήσεις μας για τα αποτελέσματα και επίσης προσπαθούμε να καταμετρήσουμε και πάλι τα αποτελέσματα των προηγουμένων σχεδίων και η Κομισιόν νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μας ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Αν όχι, παρακαλώ επαναλάβετε το ερώτημά σας. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γνωρίζω κατά πόσον οι απαντήσεις σας ικανοποιούν. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος θέλει να επανέλθει. Γιάν, ναι. ε, κάποιος μου ζήτησε να κάνω μια ερώτηση εκ μέρους του. Για την επενδυτική διευκόλυνση είναι τμήμα του ελέγχου της KPMG ή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος κάνει τον έλεγχο. Όχι, και η PMG κάνει όλους τους ελέγχους, αλλά δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο... Νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο κάνει τον επιπλέον έλεγχο αν χρειαστεί. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ωραία. Αν ε, έχει ικανοποιηθεί με τις απαντήσεις ο εισηγητής και δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάρτον. Έχουμε πολλές εκθέσεις που καλύπτουν ε, μια μεγάλη ποικιλία της δουλειάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να πω ότι η δήλωσή σας ε, ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής της διάταξης, σημείο 4, απαλλαγή 2012, άλλα όργανα. Και πληροφορήθηκα ότι ο συγητής, ο κύριος Σόνικ, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά ο κύριος Τάμας Ντόιτς είναι παρόν μεταξύ μας. και το αρμόδιο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου δεν μπορεί να είναι παρόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, για τους λόγους της εκλογής του Πρόεδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μπορούμε όμως να ακούσουμε και την άποψη των άλλων θεσμικών οργάνων, των οποίων τους εκπροσώπους χαιρετίζουμε. Μπορώ λοιπόν <clears throat> να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και εάν θέλουν να τους ζητήσω να λάβουν το λόγο. Αν θέλει ο συνεισηγητής κύριος Δόης μπορεί να λάβει το λόγο για τις προκατακτικές του παρατήρησης. Όχι. Οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ποιος είναι παρόν από την Επιτροπή των Περιφερειών. European the Okay. Ja, dann schlage ich vor, dass wir mit dem Euro Μπορούμε να περάσουμε στο γραφείο του ε- Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κύριε Χάρντεν, μπορείτε να λάβετε το λόγο εσείς. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι παρόν. Όχι, είσαστε εδώ, είσαστε, εντάξει. Εάν θέλετε να κάνετε εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, μου δίνετε το λόγο. Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Κάποιοι από εμά εδώ δεν έχουμε διερμηνία. Αυτό ήθελα να σας πω. Όσον αφορά την ε, συνέχεια μετά τις παρατηρήσεις που έγιναν ε, με την απαλλαγή του 2011, α, δεν σας είπα ποιος είναι ο συναδερφός μου εδώ, ο κύριος Γκέχαρντ Γκριλ, ο οποίος είναι ο διευθυντής, ο υπεύθυνος για δημοσιονομικά ζητήματα στην υπηρεσία του διαμεσολαβητή. Λοιπόν, επανέρχομαι στην απόφαση απαλλαγή του 2011. Στο σημείο 4 ζητούσατε να βελτιωθεί το ποσοστό χρήσης και το 2012 αυξήσαμε όντως το ποσοστό αυτό περισσότερο από τρει μονάδες και πήγε στο 95,8% σε σχέση με το 92,44% που είχαμε το 2011. Στο σημείο 9 Επίσης αναφέρεται στις προσφυγές και ζητήσατε να βελτιωθεί το ποσοστό αποφάσεων του παραδεκτού στις προσφυγές που έφταναν σε μας. Το 2012 επιφέραμε σημαντικές αλλαγές στην αρχική διαδικασία προσφυγών και η επίπτωση ήταν πολύ σημαντική, ο αντίκτυπο ήταν μεγάλο. Το ποσοστό των ε, αποφάσεων του ε, παραδεχτού πήγε στο 85% σε 18 μήνες αντί για 75% που ήταν το 2011. Ο στόχος για τον δίκτυ απόδοσης παραμένει το 90%. Και φαίνεται ότι θα φτάσουμε πιο κοντά στο 90% το 2013. Το 2012 από 70% πήγαμε στο 85%. Στο σημείο 10 του ψηφίσματος επίσης ζητάτε μείωση του όγκου των ερευνών ε, του μήκους της έκθεσής μας καταφέραμε να φτάσουμε πολύ κοντά στο στόχο μας, γιατί 77% των υποθέσεων έκλεισαν σε 12 μήνες. Πετύχαμε δηλαδή το στόχο του 69%. Θα ε, ξαναδούμε βέβαια τον ε, στόχο αυτό το 2014 και κατά πάσα πιθανότητα θα θέσουμε έναν ακόμα πιο φιλόδοξο στόχο. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 40% των περιπτώσεων για τις οποίες ζητάμε γνωμοδότηση από, την, από τα άλλα κοινοτικά όργανα, χρειάζεται περισσότερους γύρους με ρωτήσεις, με προτάσεις για μια ε, λύση φιλική. Οπότε είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις να κλείσουν υποθέσεις σε 12 μήνες. Ακόμα και αν το άλλο κοινοτικό όργανο ανταποκρίνεται στις προθεσμίες που ζητάμε εμείς. Πάντως, με την συνεργασία, με την καλή συνεργασία θα μπορούμε σε 10 μήνες να κλείσουμε κάποια υπόθεση. Σημείο 11 του ψηφίσματος. Ζητάει καλύτερη ανάλυση των πόρων προκειμένου οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε σχετική ανάλυση βάσει της οργανωτικής δομής του γραφείου του Διαμεσολαβητή. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όμως με τα αποτελέσματα γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μια που τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων ή τμήματων. Συνεπώς, εγκρίναμε μια διαφορετική προσέγγιση βασιζόμενη στη βέλτιστη πρακτική μέσω συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα λειτουργικό πλαίσιο, operating framework, business model το λένε αλλού στον ιδιωτικό τομέα, που αναλύει τις διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στην ετήσια στρατηγική του Ombudsman. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε ήδη μεταφέρει ανθρώπινους πόρους, έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες, 5% έχουν αυξηθεί οι ανθρώπινοι πόροι που ασχολούνται με τις έρευνες. Βελτιώνουμε επίσης το πλαίσιο αυτό και την επόμενη χρονιά, θα φανεί αυτό στην έκθεσή μας που θα είναι του Μαρτίου, και αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το προσωπικό. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάρτον. Σας, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντέ, Διευθυντά. Βλέπω τώρα βλέπω το, σχέδιο το οποίο είχαμε ενώπιον μας. Έχουμε ζητήσει από όλα τα θεσμικά όργανα να ακούσουμε τις απόψεις τους και μετά στο τέλος το προβλεπόταν το ελεγκτικό συνέδριο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 Εκτελώ Γενικού ε, Γραμματέα, ο κύριος Φρέντ είναι δίπλα μου, ε, που είναι Διευθυντής ε, Προϋπολογισμού και Οικονομικών να σας μιλήσω για το διορισμό του νέου ε, Γενικού Γραμματέα που έχει δρομολογηθεί εδώ και μερικούς μήνες ε, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχω κάποιες ε, δηλώσεις να κάνω. Καταρχάς, η ΟΚΕ πάντοτε ήταν ιδιαίτερα διαφανής στα ανώτατα επίπεδα διαχείρισής της. Το βλέπετε και στην ετήσια έκθεση που μεταξύ άλλων ε, συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα του εκτονιστέρων ε, ελέγχου. Δεύτερον, ε, επικροτούμε τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του το 2012 για, κατά στο πλαίσιο της οποίας δεν υπήρξαν, δεν εμφανίστηκαν σφάλματα για την ΕΟΚΕ. Χαίρομαι λοιπόν ε, που βλέπω ότι το πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η ΕΟΚΕ δουλεύει πολύ καλά. Να τονίσω επίσης τη σημασία της ε, της ε, Συμφωνίας Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ξέρετε ότι είναι παλιά συμφωνία, δεν είναι καινούρια. Είναι όμως σημαντικό να τονίσει κανείς τη σημασία της. Η τρέχουσα συμφωνία εκπνέει στα τέλη του τρέχοντος έτους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και ε, πρέπει να ανανεωθεί. Έχουν αρχίσει οι σχετικές συνομιλίες με την Επιτροπή των Περιφερειών. Η συμφωνία ε, σημαίνει πολλά ωφέλη ε, ως προς τη συνεργασία και είναι πραγματικά μοναδική μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θέσω αφορά τη Συμφωνία Συνεργασίας και τις σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής ε, Περιφερειών ε, και της Οικονομικής και Κοινωνικής ε, Επιτροπής και από την άλλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια συμφωνία με ένα πολιτικό τμήμα και ένα διοικητικό τμήμα. Ε, αναμένω εναγωνίως ε, να δω αμοιβαία ωφέλη αυτής της ε, συνεργασίας. Ξέρετε ότι έχει εγκριθεί από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αρχές Δεκεμβρίου και τώρα επαφίεται την επόμενη εβδομάδα στην, στο Προεδρείο της ε, ε, ΕΟΚΕ την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη της Επιτροπής Περιφερειών να, να εγκρίνουν αυτή τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καλύπτει και πολιτικές και διοικητικές πτυχές. Όπως γνωρίζετε υπάρχει πρόβλεψη ε, συγχώνευσης με την μεταφραστική υπηρεσία ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και τη δημιουργία ενός νέου τμήματος έρευνας. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους κανόνες αποζημίωσης των μελών κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ενέκρινε το, την ε, εκτελεστική απόφαση το Νοέμβριο, και τα νέα, τα νέα, οι νέοι κανόνες για την αποζημίωση των μελών εφαρμόζονται ήδη από 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτά ε, από μέρους μου για την ώρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αλεξόπουλο. Και στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κόλια από το ελεκτικό συνέδριο. Έχετε το λόγο. Sorry. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. Σας ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο. Το 2012 ήταν πολύ σημαντικό έτος για το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, ήταν η περάτωση της στρατηγικής του το 2005-2012 και υλοποιήθηκαν τα περισσότερα αποτελέσματα τα οποία ε, έπρεπε να είχαν επιτευχθεί μέχρι τότε. Κύρια επιτεύγματα. Πετύχαμε μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των των εκθέσεών μας και ποσοτικά και σε ποιότητα αυξήθηκε και η εκτίμηση για την ποιότητα αυτών των εκθέσεων από τους κύριους εμπλεκομένους και υπήρξε και μεγαλύτερο επίπεδο αποδοχής των συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου από την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση πόρων στο ελεκτικό συνέδριο, υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε αποτελεσματικότητα, για να σας δώσω δύο παραδείγματα. 40 μέλη του προσωπικού περάσαν από διοικητικές υπηρεσίες <clears throat> σε υπηρεσίες ελέγχου. Επίσης δημιουργήσαμε ένα σημαντικό νέο κτίριο για το ελεκτικό συνέδριο. Πέραν από την εξοικονόμηση για τα μισθώματα, συνενώνει όλες τις υπηρεσίες μας κάτω από, τον ίδιο, κάτω από την ίδια στέγη και βοηθάει την αποτελεσματικότητα του ελεκτικού συνέδριου. Για το 2012 ιδιαίτερα. Ήταν η χρονιά που το ελεκτικό συνέδριο εστίασε στο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προετήθει για τις σημαντικές ε, προκλήσεις του 2013 και επέκεινα. Εγκρίναμε λοιπόν 10 γνωμοδοτήσεις και άλλα έγγραφα <clears throat> για κυρία πακέτα προτάσεων νέων κανονισμών όπως αυτό αφορά την ε, έρευνα και καινοτομία με τον ορίζοντα 2020, τη γεωργία και άλλα. Το 2012 ήταν και ένα έτος φτάσαμε το επίπεδο 25 σε σχέση με το έτος που δημιουργήθηκε στρατηγική που ήμασταν στο επίπεδο 12. Τα, οι εκθέσεις μας για τους αποκεντρωμένους φορείς έφτασε στο επίπεδο των 50 εκθέσεων έναντι 29 το 2008. Και επιπλέον, πρόκειται για ένα έτος όπου η ποικιλία των ε, <clears throat> θεμάτων που αντιμετωπίσαμε ήταν χωρίς προηγούμενο. Αντιμετωπίσαμε θέματα όπως τα σχέδια αποδοτικότητας ενέργειας, ε, λιμενικές εγκαταστάσεις, αποτελεσματικότητα στα σφαγεία και το Ταμείο Προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι τώρα το έργο ε, λογιστικού ελέγχου που γίνεται από το ελεγκτικό συνέδριο προς την κατεύθυνση ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Έχουμε 565 ελεγκτές οι οποίοι εργάζονται στο Λουξεμβούργο και επιτοπίως και το 2012 κάναμε 6.816 μέρες ε, επιτόπιων ερευνών και ένα μεγάλο μέρος των οποίων ήταν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου, 98% από αυτές έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν και 80% από αυτές έχουν εφαρμοστεί, για να δείτε ποιος είναι ο αντίκτυπος του έργου μας. Για το επίκαιρο των εκθέσεών μας έχουμε κάνει σημαντικές βελτιώσεις στο χρονικό αυτό διάστημα για την χρονική στέρηση που χρειάζεται ώστε να εκδοθεί μια έκθεση. Έχουμε φτάσει το 2012 σε 20 μήνες, ενώ <clears throat> το 2008 ήταν 25 μήνες κατά μέσον όρο, αλλά παρόλα αυτά το ελεκτικό συνέδριο προσπαθεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα έκδοσης αυτών των εκθέσεων. Γι' αυτό τονίζουμε ότι αυτός ο τομέας είναι μια κέρια προτεραιότητα στην στρατηγική μας για το 2013 με 2017. Τέλος, στο τομέα της διαχείρισης των πόρων, θέλω να σας αναφερθώ σε τρεις περιοχές. Πρώτα απ' όλα, το 2012 πετύχαμε σημαντικό επίπεδο απορρόφηση των κονδυλίων 96% και μόνο 3% και νέες θέσεις. Δεύτερον, τον Οκτώβριο του 2012 περατώσαμε το νέο μας κτίριο και είναι το κτίριο όπου βρισκόνται οι ελεκτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφορικής του ελεκτικού συνεδρίου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα μετά από την περάτωση του κτηρίου χρειάστηκε να μεταφέρουμε όλο το κέντρο δεδομένων του ελεκτικού συνεδρίου. Ήταν δύσκολο εγχείρημα αλλά πέρασε πολύ. Τρίτον, έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε τις περισσότερες από τις συστάσεις του εσωτερικού ελεκτή του ελεκτικού συνεδρίου και επίσης και τις ε, συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή, αυτό δείχνει την ευρωστία των εσωτερικών συστηματών ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου. Κατά τα άλλα, με στη διαθεσή σας να απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε ίσως θέση. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Κόλια, λέει ο πρόεδρος για την εκθεσή σας από το ελεκτικό συνέδριο. Και τώρα στρέφομαι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Γενικό Διευθυντή, κύριο Ουμής. Euh, Ευχαριστώ. Ναι, είμαι Γενικός Διευθυντής Προσωπικού και Δημοσιονομικών στο Ελεκτικό Συνέδριο, στο, συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας κατά το 2012. Συγχρόνως ζητούμε συγγνώμη τον υπεύθυνο του δικαστηρίου που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, τον ε, γραμματέα μας δηλαδή. Πάντα ήταν επιστός αυτό το ετήσιο ραντεβού με την Επιτροπή σας, γιατί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις συστάσεις σας κάθε φορά που παρουσιάζετε εκθέσεις για την απαλλαγή. Θα διαπιστώσατε μάλιστα ότι και σε άλλες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του 2012 λαμβάνουμε υπόψη μας τις συστάσεις που γίνονται σε σχέση με την απαλλαγή 2011. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής τη άσκησης διαφάνειας, την οποία έχουμε σήμερα, θέλω να αναφερθώ κυρίως σε δύο ζητήματα αφενός στην χρήση των πόρων, πώς χρησιμοποιούμε δηλαδή τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από τη Δημοσιονομική Αρχή και δεύτερον στην ε, δραστηριότητα την ομολογική του δικαστηρίου μας. Όσον αφορά τους πόρους, πολύ σύντομα. Εδώ θα έλεγα ότι η ανησυχία μας είναι να χρησιμοποιούμε τους πόρους όσο γίνεται καλύτερα είτε πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό, είτε πρόκειται για οικονομικούς πόρους. Θέλουμε λοιπόν μια βέλτιστη χρήση και ποσοτικά, μια που έχουμε ένα ποσοστό χρήσης των κονδυλίων που είναι της τάξεως του 99% και όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης 98% περίπου. Θέλουμε επίσης βέλτιστη χρήση και ποιοτικά διαπιστώνουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 δεν διατύπωσε καμία παρατήρηση όσον αφορά την διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλά το σύστημα ελέγχου μας και δεν διαπίστωσε καμία παρατυπία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους πόρους. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο. Θα αναφερθώ λιγάκι Έρχομαι τώρα λοιπόν στις δραστηριότητες που αφορούν τη δικαιοδοσία του σώματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ελέγχει το φόρτο εργασίας του πρώτα απ' όλα. Οι διάφορες υποθέσεις φτάνουν στο δικαστήριο και το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τις υποθέσεις αυτές, να επιλέξει κάποιες, να μην ασχοληθεί με άλλες κλπ. Πρέπει να ασχοληθεί με όλες τις υποθέσεις που φτάνουν σε αυτό βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται. Εξάλλου, ο φόρτος αυτός εργασίας αυξάνει συνεχώς. Τα πέντε τελευταία χρόνια οι υποθέσεις που μας έφτασαν αυξήθηκαν πάνω από 20% και που εξετάστηκαν από εμά, κάθε χρόνο έχουμε 5% αύξηση. Το 2012 είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια μικρή μείωση. Η μείωση όμως αυτή ήταν προσωρινή. Το 2013 είχαμε και πάλι ε, μεγάλη αύξηση της ε, τάξης του 10% και παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό δυστυχώς σημαίνει αύξηση των υποθέσεων που παραμένουν σε κρεμότητα. Και τα διάφορα ζητήματα που ετέθησαν κατά τη διάρκεια της ε, απαλλαγής, πολλά αναφέρονται ακριβώς αυτό το θέμα των υποθέσεων σε κρεμότητα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά. Γι' αυτό και το Δικαστήριο τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε διάφορα μέτρα, μικρά, μεγάλα, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, ώστε η αύξηση αυτή των υποθέσεων να μην καταλήγει σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες. Επίσης θέλουμε όσο γίνονται περισσότερες υποθέσεις να τις ευεξεργαζόμαστε και να τις τελειώνουμε. Πήραμε λοιπόν πολλά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα νομοθετικά μέτρα, ρυθμιστικά μέτρα, ε, μεταρρύθμιση δηλαδή του καταστατικού του δικαστηρίου και μεταρρύθμιση του κανονισμού όσον αφορά τις ε, διαδικασίες σε σχέση με τη δικαιοδοσία μας. Υπήρξε για παράδειγμα αύξηση του αριθμού των ε, τμήματων που κρίνουν τις υποθέσεις. Επίσης είχαμε έναν παραπάνω γενικό εισαγγελέα ο οποίος μας ήρθε τον Οκτώβριο που μας πέρασε και δύο άλλοι θα μας έρθουν το 2015. Απλοποίησαμε επίσης τις διαδικασίες. Έχουμε τη δυνατότητα να ε, εξετάζονται πιο γρήγορα υποθέσεις χωρίς ακρόαση και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο σχέδιο που λέει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών. Κάναμε σχετική πρόταση στις νομοθετικές αρχές. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε, η Επιτροπή Προπολογισμών επίσης. Δυστυχώς όμως η πρόταση αυτή βρίσκεται στο Συμβούλιο και εκεί έχει κολλήσει γιατί οι εθνικές αντιπροσωπείες δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τον αριθμό τελικά των επιπλέον δικαστών και για τον τρόπο με τον οποίο θορίζονται αυτοί. Και είναι κρίμα γιατί και πάλι ε, υπάρχει συμφόρηση στο δικαστήριο. Ενώ θέλουμε να μπορούμε να δουλεύουμε πιο γρήγορα. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα. Δεύτερα, δεύτερη κατηγορία μέτρων. Ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης που έχουν να κάνουν με επεξεργασία θεμάτων δικαιοδοσίας. Η Δημοσιονομική Αρχή συμφώνησε το 2013 προκειμένου να αλλάξουν θέσεις που είχαν να κάνουν με βοηθούς και να αντικατασταθούν από νομικούς, ώστε να ενισχυθεί έτσι η δυνατότητα διαχείρισης υποθέσεων των γραφείων των δικαστών. Επίσης, δημιουργήθηκε και ένα επιπλέον γραφείο Γενικού Εισαγγελέα του 2013 και όσον αφορά τον προπολισμό του 2014 πετύχαμε την ε, δημιουργία νέων ε, θέσεων επιπλέον στο δικαστήριο κάτι το οποίο αντισταθμίζει κατά κάποιο τρόπο την απουσία ε, της ε, προσθήκης 12 δικαστών που όπως ε, σας είπα έχουμε ζητήσει. Λοιπόν, οι θέσεις αυτές ασχολούνται με τις υποθέσεις του μας, βέβαια χωρίς να προκαταλάβουμε και Τόσα όσα μας επιβάλλονται από τη Δημοσιονομική Αρχή για μείωση 1% κάθε χρόνο του προσωπικού μας για τα επόμενα χρόνια. Και έχουμε ήδη μείωση κατά 20 της απασχόλησης το 2013 και 20 το 2014. Αλλά έχει να κάνει περισσότερο με θέσεις απασχόλησης της υπηρεσίας. χωρίς ε, να πληγεί ενίσχυση του προσωπικού μας στην επεξεργασία των υποθέσεων. Και θα προσθέσω και ένα τρίτο θέμα για τα μέτρα που υιοθέτησε το δικαστήριο για να είναι πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό και αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη περισσότερων ε, εργαλείων πληροφορικής. Γίνεται μία προσπάθεια με το σύστημα e που επιτρέπει ηλεκτρονικά ε, μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στις ε, διάφορες πλευρές, δηλαδή κατάργηση του χαρτιού όσο γίνεται. Όπως επίσης και μέσω ηλεκτρονικών αρχείων για την ε, νομολογία που σημαίνει ότι χιλιάδες σελίδες χαρτί καταργούνται. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα στοιχεία που είχα να σας μεταφέρω. Τέλος, επιτρέψτε μου να προσθέσω δύο λόγια. Διαπιστώνουμε ότι είχαμε πάντα μεγάλη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Νομική Επιτροπή και εκείνη των προπολογισμών, προκειμένου να μας δοθούν τα μέσα που ζητάμε για να ενισχυθεί η ικανότητά μας, η ικανότητά μας κρίσης των διαφόρων υποθέσεων που μας φτάνουν. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας αυτή, για την κατανόησή σας και ελπίζω με την παρέμβασή μου να σας βοήθησα να καταλάβετε καλύτερα το τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ό,τι ερωτήσεις έχετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, ο κύριος Στάλνας, που είναι Γενικός Γραμματέας τη Επιτροπής των Περιφερειών. Ήρθε. Πού είσαστε? Α, εκεί. Ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας μιλήσω για τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών και να απαντήσω και στον κύριο Λεμπράν, τον εισηγητή και πρόεδρο της Επιτροπής μας ε, ΚΑΦΕΚ που είναι επίσης εδώ. Ευχαρίστω στη συνέχεια να απαντήσουμε και σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Το 2012 ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή των Περιφερειών και η πολιτική μας εργασία ενισχύθηκε ιδιαίτερα, αλλά και υπήρξε βελτίωση της αποδοτικότητας της διοικητικής δομής της Επιτροπής των Περιφερειών. Να σας δώσω μονάχα ορισμένα στοιχεία για το πολιτικό έργο της Επιτροπής των Περιφερειών ως υπόβαθρο για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα πώς χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι της διοίκησης. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει βελτιώσει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι υπήρχε μεγαλύτερη συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πολιτικό έργο της Επιτροπής των Περιφερειών. Υπήρξαν κοινέ συναντήσεις με την, ε, με, τις Επιτροπ... Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου <clears throat> και συνεργασία για την προετοιμασία του κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων και επίσης μια πολύ στενή συνεργασία με επαφή μεταξύ εισηγητών και επιτροπών. Επίσης το θέμα των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Περιφερειών και υπήρξε συνεργασία του εισηγητή μας με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ίδια αυτά θέματα. Έχουμε επίσης αναπτύξει και ένα δίκτυο σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά και φυσικά και εδώ υπήρξε στενή συνεργασία με άλλα ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω τα νομοθετικά όργανα σε ό,τι αφορά και τα θέματα της ε, αναδυόμενης οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Επιτροπή των Περιφερειών αντιμετώπισε το θέμα της επικορικότητας και της εφιούς ε, ρύθμισης με συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των αρχών που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα. Τη συμπερίληψή του λοιπόν στο συνολικό νομοθετικό αργό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης υπήρξε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαδοχικών προεδριών υπήρξε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο οδήγησε στην έκδοση γνωμοδοτήσεων ετής του Συμβουλίου από την Επιτροπή των Περιφερειών για θέματα τα οποία θεωρήθηκαν σημαντικά από το Συμβούλιο. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε να κατανοήσετε γιατί η Επιτροπή ε, των Περιφερειών κατάφερε να χρησιμοποιήσει τους περιορισμένους τους πόρους επιτυχώς το 2012 για να μπορέσει να ενισχύσει αυτές τις ε, ενέργειες. Η Επιτροπή των Περιφερειών έκανε μια σημαντική προσπάθεια για να συνεχίσει τη βελτίωση της, ε, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του διοικητικού του μηχανισμού. Ήδη σε προηγούμενες ε, διαδικασίες απαλλαγής έχει κατανοήσει η Επιτροπή σας ότι εμείς προχωρούμε στην διαδικασία της ε, Επιτροπής των Περιφερειών στο, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά θέματα με τη διαδικασία ΚΑΦ ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αποτελεσματικότητα. με την προσπάθεια αυτή βελτίωσης της χρήση των ανθρωπίνων πόρων, η Επιτροπή των Περιφερειών ακολούθησε τον κανόνα ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να μειώσουν κατά 2% το κόστος τους με αντίστοιχη αύξηση της ε, αποτελεσματικότητας και μόνο τότε μπορούν να τους δοθούν προσωπικό εάν επιτύχουν αυτό το 2% εκτός αν είναι μια σημαντική προτεραιότητα πολιτικού χαρακτήρα η οποία απαιτεί περισσότερο προσωπικό. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού μας υπήρξε φυσικά η αβεβαιότητα η οποία μας ταλάνισε σε ό,τι αφορά τα θέματα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ε, ε μισθών γιατί 55%, από το, τις δαπάνες μας συνδέονται με κόστος προσωπικού και επομένως ήταν πολύ σημαντικότερη η ανασφάλεια που αντιμετωπίσαμε από άλλα όργανα διότι συνδεόταν με τα μισθολογικά επίπεδα. Παρόλα αυτά και μόνον τούτο η Επιτροπή των Περιφερειών μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο κατάφερε να εξασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό της. Και με τα περιορισμένα μέσα που έχουμε λοιπόν και με ένα ε, όργανο το οποίο είναι σχετικά νέο, <clears throat> έχουμε βελτιώσει την διοικητική μας ικανότητα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο αυτό και φυσικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ενισχύσουμε τη διαθεσμική συνεργασία Είχαμε τη συνεργασία σε διοικητικό επίπεδο με την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες και προσπαθούμε να καταλήξουμε και σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα σε ό,τι αφορά την πολυγλωσία. Το Προεδρείο μας αποφάσισε ότι η διαδικασία μετάφρασης θα ε, πρέπει να αναδιαφθορθεί ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μετάφρασης και έτσι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια μορφή πολυγλωσσίας που είναι αποτελεσματική σε σχέση με τη χρήση των πόρων και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ε, μεταφραστικές μας ε, ικανότητες, κάτι που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας για να καλύψουμε νέους τομείς δραστηριότητες και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η διαθεσμική συνεργασία, το να ενισχυθεί περισσότερο και στα θέματα αυτά οι πολιτικές μας αρχές έχουν ε, τονίσει τη θέλησή τους να ενισχυθεί ακόμα περισσότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να μπορέσει να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάλ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της συζήτησης. Και έχουμε επίσης και ένα ακόμα θεσμικό όργανο που είναι ο επόπτης προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Ντόξη, τον διευθυντή του φορέα αυτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μαριάν Σάντσες Λόπεζ είναι εδώ, υπεύθυνη οικονομικών ε, του οργανισμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε για να σας πούμε τι κάνουμε ε, τον τελευταίο χρόνο. Εγώ δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Προστασίας ε, των Δεδομένων. Είμαστε το νεότερο όργανο. Την επόμενη εβδομάδα θα γιορτάσουμε τα δέκατα γενέθλιά μας. Ελπίζουμε να μας... Ελπίζουμε να γιορτάσετε μαζί, μαζί μας. Κάθε φορά που γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικών σας αλλά και όλων των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχουν σχετικοί νόμοι που προστατεύουν την ε, επεξεργασία των δεδομένων αυτών εγκρίναμε μια στρατηγική για το 2013-2014 για να λάβουμε υπόψη ε, την πρόκληση της αύξησης ε, των δραστηριοτήτων μας και της διεύρυνσης αυτών. Ε, κάναμε και σχετική έκθεση για το θέμα αυτό. Την επόμενη χρονιά θα είναι πιο λεπτομερής η έκθεσή μας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην συνέχιση των συστάσεων και των παρατηρήσεών σας σε σχέση με την απαλλαγή για το 2011. Σε σχέση με τη σύσταση παριθμών 5, το 2009 το ελεγκτικό συνέδριο συνέστησε να βελτιώσουμε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ε, εγγράφων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των υπαλλήλων. Εμείς ε, βελτιώσαμε την ε, κατάσταση το 2010 και το 2010 μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι κάναμε κάποια πράγματα για την βελτίωση ε, την, της ε, κατάστασης και μάλιστα μας είπε ότι δεν υπήρξαν σφάλματα για τη χρονιά αυτή. Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού μας σε σχέση με ε, τις επιστώσεις υποχρεώσεων έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. 95,1% 95, ε, το 2012, ενώ ήταν 89,1% το 2011 για τα σημεία 7 και 8. Η εκτέλεση του προπολογισμού σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών επίσης βελτιώθηκε η ε, κατάσταση και βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα αυτό ήταν ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός νέου δημοσιονομικού εργαλείου που χρησιμοποιήσαμε το 2011 και από 85,03% το 2011 φτάσαμε σε 89,69% το 2012 ως προς την εκτέλεση των πληρωμών. Για το σημείο 12 τώρα, των παρατηρήσεων ε, εγκρίναμε τη στρατηγική για το 2013 και 2014 πέρυσι με σύνολο στόχων, δράσεων και βασικών ε, δικτών επιδόσεων για να παρακολουθήσουμε καλύτερα τη δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας σε σχέση με τη χρήση των πόρων και θα ήθελα να τονίσω ότι μας βοήθησε και μας συμβούλευσε πάρα πολύ το ε, ελεγκτικό ε, συνέδριο αλλά και το γραφείο του διαμεσολαβητή γιατί είδαμε ε, πόσο πολύ είχαν χρησιμοποιήσει αυτούς τους δείκτες ε, επιδόσεων για ε, την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Έχουμε φτάσει στο 90,3% για την εκτέλεση φέτος ήδη. Θα είχαμε φτάσει ε, ίσως ακόμη, και υψηλότερα κατόπιν ε, των συστάσεων ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Ελπίζουμε να φτάσουμε ακόμη ε, σε ακόμη ψηλότερο ποσοστό. Έχουμε επίσης και ένα σύστημα διαχείρισης συγκεκριμένων περιπτώσεων. Μας πήρε λίγο χρόνο βέβαια να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες και τις ασφάλειες, τις εγγυήσεις για την ασφάλεια του συστήματος. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις και αυτή τη στιγμή το καταφέραμε έχουμε τώρα ε, περάσει στη χρήση του συστήματος που είναι πλέον πλήρως λειτουργικό. Και τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τη δήλωση αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2012, τη λεγόμενη DAS, το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχε παρατηρήσεις ε, κατόπιν του ελέγχου του σε σχέση με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών μας και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντόξη. Τέλος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή ε, ΚΡΙΣΠ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού ε, Συνεδρίου. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας εύχομαι Καλή και ευτυχισμένη χρονιά 2014 εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ζητώ συγγνώμη που δεν είναι κανένας άλλος. Από εκεί έχουμε δύο διευθυντές και διάφορους άλλους ε, από το τμήμα μας. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι η εικόνα είναι πολύ ωραία, γιατί το επίπεδο σφάλματος είναι μηδενικό Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία έκθεση για σας. Πάντως, υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές στην προσέγγιση μας φέτος. Η πρώτη έχει να κάνει με μια αλλαγή στην αναρμόνιση της πολιτικής, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα των αναθέσεων. Πρώτα απ' όλο, ο τομέας των διοικητικών δαπανών ενέχει ναι, ναι, χαμηλό επίπεδο κινδύνων Με την αλλαγή στην ε, μεθοδολογία για την εκτίμηση σφάλματος στις δημόσιες συμβάσει, ε, είδαμε ότι αν εντοπίζεται ένα τέτοιο λάθος, τότε αμέσω μπαίνει στους λογαριασμούς. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε συνετοί και να αυξήσουμε τον αριθμό των δειγμάτων ε, κατά τρία, προκειμένου να υπάρξει ένα περιθώριο αν θέλουμε να βρούμε κάποιο σφάλμα και έτσι να μπορούμε να σας δώσουμε κάποια ασφάλεια για τις δαπάνες στο τομέα αυτό. Οι δαπάνες έχουν να κάνουν κυρίως με τους μισθούς, τις ε, συντάξεις, κτίρια, πληροφορική. Δεν βρήκαμε κανένα σφάλμα όσον αφορά τις συμβάσεις. Οι μόνες αδυναμίες έχουν να κάνουν με τα συστήματα. Και έτσι έρχομαι στη δεύτερη μεθοδολογική μας τροποποίηση. Αποφασίσαμε ότι αφού δεν μπορούμε κάθε χρόνο να εξετάσουμε όλα τα συστήματα, θα γίνεται εκ περιτροπής. Αν θεσμικό όργανο και την συγκεκριμένη χρονιά πήραμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εξετάσαμε συστήματα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές είναι θετικά τα αποτελέσματα. Καταλήξαμε ότι οι διάφορες συναλλαγές που έχουν να κάνουν διοικητικές δαπάνες το 2012 δεν έχουν σφάλματα, κρίνονται ε, κανονικές, διοπιστώνονται κάποιες ε, αδυναμίες στο σύστημα και στις κοινωνικές παροχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους εισηγητές εξ των θεσμικών οργάνων και μετά από τον ε, εισηγητή του Ελεκτικού Συνεδρίου θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάμας Ντόις, τον συνεισηγητή για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε και ο, ο πρόεδρος μας στις ε, αρχικές του παρατήρησης, πρόκειται για την πρώτη μας ε, συνεδρίαση το 2014. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και να όλους που είναι παρόντες από τα διάφορα θεσμικά όργανα και να ευχηθώ σε όλους και στους συναδέλφους μου επίσης καλή χρονιά. Για το σημείο αυτό τώρα της ημερησίας διάταξης που είναι η απαλλαγή των θεσμικών οργάνων για το 2012 θα ήθελα και εξ του συναδέρφου μου του Μπόγουσλα Σόνικ να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει ε, για, το, για το έργο αυτό το ελεκτικό. Το 2012 και η απαλλαγή που συνδέεται με το έτος 2012 είναι η βάση για την έκθεση την οποία έχουμε συντάξει μαζί με τον κύριο Σόνικ. Ο στόχος μας ήταν να αντιμετωπίσουμε την απαλλαγή του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό σε μία σειρά συζητήσεων. και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε προβλήματα τα οποία να έχουν αναδειχθεί για τα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Πήραμε πλήρες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μας, έχουμε επεξεργαστεί αυτά τα ερωτηματολόγια και παρά το γεγονός ότι κάποιες απαντήσεις μπορεί να δώσουν λαβή σε περαιτέρω ερωτήσεις, νομίζω ότι έχουμε μια σαφή δομή στη συζήτησή μας και έχουμε κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχαμε θέσει το ερώτημα των περιπτώσεων που ήταν ακόμα εκκρεμείς, των ε, δικαστικών υποθέσεων που ήταν ακόμα εκκρεμείς και μας ενδιέφερε το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα του προϋπολογισμού και πόσο αποτελεσματική ήταν η εργασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Πώς λοιπόν μπορεί με καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσει τον Ευρωπαίο πολίτη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας έδωσε τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας σχετικά. Ξέρουμε ότι εδώ και 20 χρόνια αυξάνει ο όγκος εργασίας και οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν και έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης αυτού του φόρτου εργασίας που παραμένει εκκρεμής. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα διορισμού περαιτέρων δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένω, το ερώτημα μα ήταν με ποιο τρόπο μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κάνει τι απαραίτητε ενέργειε <clears throat> ώστε να μην αυξηθεί αυτό ο φόρτο εργασία του παρελθόντο και να μπορέσει <clears throat> να ε, τύχει επεξεργασία. Το δεύτερο ερώτημα προ το <clears throat> Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το θέμα της ε, χρήσης πόρων για μετάφραση και διερμηνία για την πολυγλωσία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 2.000 εργαζόμενους και περίπου το ίμεση από αυτούς εργάζονται στους τομείς ε, μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού και φυσικά και ένα μεγάλο μέρος των δαπανών. Ποια είναι τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα αυτό για να μειωθεί το κόστος της πολυγλωσσίας στο δικαστήριο, χωρίς φυσικά αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην χρήση της πολυγλωσσίας. Και ένα ακόμα ερώτημα ήταν το θέμα της ε, διαδικασίας που έγινε από την όλα εναντίον ενός ε, υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ποια είναι η κατάσταση αυτής της διαδικασίας στην ΟΛΑΦ ήταν το ερώτημα. Έρχομαι τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. Είχαμε τα δύο ερωτήματα αυτά που ήταν ίδια και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παραγωγός χάρη, ποιο είναι το κόστος της πολυγλωσσίας το κόστος μετάφρασης, και όπως αναφέρθηκε από τα δύο όργανα κοστίζει στο ένα όργανο η μονάδα μετάφρασης 98 ευρώ, στο άλλο περίπου 250 δεν θα ήθελα όμως να επαναλάβω αυτό το ερώτημα γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στο μέσο κόστος της μετάφρασης μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να γνωρίσουμε λοιπόν γιατί υπάρχει τόσο υψηλό κόστος μετάφρασης. Και ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε μια τόσο μεγάλη διαφορά. Ίσως είναι ένα θέμα μεθόδου Καταμέτρηση του κόστου, αλλά σαφώ υπάρχει μία διαφορά. Και σε ό,τι αφορά την Όλαφ, πήραμε την απάντηση ότι υπάρχει μία διαδικασία της Όλαφ εναντίον ενός συνεργάτη του ελεκτικού συνεδρίου και εδώ το ερώτημα μας φυσικά ήταν σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η διαδικασία και αν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία. το 2012 το ελεκτικό συνέδριο είχε 16 πιθανές περιπτώσεις απάτης ε, διαβιβάσεις στην ΟΛΑΦ και υπήρξαν εσωτερικές διαδικασίες στο ελεκτικό συνέδριο για αυτές τις 16 υποθέσεις. Σε 9 περιπτώσεις η ΟΛΑΦ ξεκίνησε έρευνες. Μήπως θα μπορούσε να μας πει κάτι περισσότερο για το θέμα αυτό το ελεκτικό συνέδριο ήταν το ερώτημά μας. Και θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι και τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών. Τέλος. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ κάπως εκπληκτικό το ελεγκτικό συνέδριο έκανε 24 συναντήσεις όπου έπρεπε να είναι παρόντα όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά μόνο σε μία από αυτές ήταν παρόντα όλα τα μέλη του συνεδρίου. Επομένως υπάρχει το πρόβλημα αυτό απουσιών. Το ερώτημά μου, αν οι εσωτερικοί κανόνες του ελεκτικού συνεδρίου προβλέπουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αν κατά πόσο έχουν τηρηθεί. Και γιατί υπήρξε μια τόσο μεγάλη έλλειψη παρουσίας των μελών του ελεκτικού συναδρίου. Υπήρξε μοναχαμία περίπτωση που ήταν παρόντα όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Και το, αυτά ήταν τα ερωτήματα μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε. και θα χαιρόμουν να ακούσω και τις, απαντήσεις, ερωτήσεις άλλων συναδέλφων καθώς και απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ντόιτς. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να θέσει κάποια ερωτήματα. Η κυρία Γκρέσλε, ο κύριος Γκάιερ. Κυρία Γκρέσλε. Λυπάμαι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχήν που δεν μπόρεσα να είμαι στην αρχή της συνεδρίασης. Έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Βιομηχανίας και επίση δεν θα μπορέσω να, περιμένω όλες τις ε, απαντήσεις αλλά θα τα καταγράψει ο συνεργάτης μου. Θέλω να στραφώ στον εκπρόσωπο του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είδατε ότι είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία διατυπώσαμε σε εσά, γιατί είδαμε ότι το μήκος των ε, δικαστικών δικασιών είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί ερωτήματα και υπήρξαν και θέματα που έχουν να κάνουν με παράπονα σε σχέση με την ε, ε, απονομή διαδικασίας από χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία κτλ. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρξαν και παράπονα για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει απαραίτητη πρόνοια τους επόμενους μήνες ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο βραχία διαδικασία. στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας έχει 5.600 υποθέσεις με πολύ μικρότερο προσωπικό από ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακόμα και με τις περιπτώσεις που δεν γίνονται δεκτές από το ως παραδεκτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι, οι υποθέσεις. Είναι απαραίτητο να υπάρξει έλεγχος, να υπάρξει ε, επεξεργασία για το τι θα γίνει δεν θα γίνει ή όχι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κλείσει 55 περιπτώσεις και έχει μια μικρότερη παραγωγικότητα. Επομένως μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο μέρος του χρόνου, 15 εβδομάδες που δεν γίνεται τίποτα, δεν συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα έπρεπε να ξέρουμε λοιπόν γιατί υπάρχουν τόσες πολλές λευκές εβδομάδες μέσα στο χρόνο όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό υποθέσεων που εκκρεμούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, χωρίς μια δικαιοσύνη η οποία λειτουργεί σωστά, δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά να τονίσω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί λοιπόν υπάρχουν τόσες πολλές λευκές εβδομάδες, είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, και πόσο διαρκεί μια μέση υπόθεση από την υποβολή της μέχρι την τελική απόφαση. Και αυτό αφορά και το δικαστήριο για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα λοιπόν να έχω μία απάντηση, ενδεχομένως γραπτός, αν δεν μπορείτε τώρα να απαντήσετε αμέσως. Είπατε επίσης ότι υπάρχει αυτή η μεταρρύθμιση το 2012. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το τέλος του 2013 που βρισκόμαστε τώρα μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτής της ε, μεταρρύθμισης. Θα ήθελα και στη συνέχεια να μάθω πόσο έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία αλλά θα ήθελα να, να σας τονίσω και πάλι ότι η διάρκεια των νομικών διαδικασιών, των δικαστικών διαδικασιών θέτει σε κίνδυνο την λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. <coughs> ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ο Γιένς Γκάιερ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω όχι τόσο ερωτήσεις προς τα μέλη αυτά, αλλά περισσότερο μια αίτηση προς την Επιτροπή μας. Στην Επιτροπή μας η, η παράδοση είναι ότι ο εισηγητής συμπεριλαμβάνει τις ερωτήσεις των συναδέλφων στα δικά του ερωτήματα. Όταν δω όμως αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν απευθυνθεί στην Επιτροπή Περιφερειών και στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τις εξοικονομήσεις, αναρωτιέμαι <clears throat> αν θα έπρεπε να συμφωνήσουμε ότι ερωτήσεις αυτού του είδους δεν έχουν καμία επίπτωση στη διαδικασία απαλλαγής και θα πρέπει στο μέλλον να μην αναφέρονται. Αν κάποιος θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υπάρχει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει ό,τι η άποψή του. Αλλά όταν εμείς προχωρούμε σε μια, σε μια διαδικασία που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στη διαδικασία απαλλαγής δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να φέρνει κανείς τις προκαταλήψεις του σε σχέση με την ύπαρξη ορισμένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Εμάς μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτών των οργάνων και δεν πρέπει να αναλάβουμε μια ευθύνη για την ύπαρξη ορισμένων οργάνων που προβλέπονται ήδη από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω στους συντονιστές ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε να υπάρχει ένας περιορισμός στα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη διαδικασία απαλλαγής. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο που θέλω να θέσω. Και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο. Στο παρελθόν δεν έχουμε απασχοληθεί πάρα πολύ με το όργανο αυτό γιατί δεν ήταν τόσο αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Δεν έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα που κατονόμασε ο Τάμας Ντόιτς προηγουμένως. για διαδικασίες που υπήρξαν ε, μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και των συνεργατών τους. Θέματα που δεν εμπλέκουν μονάχα τις ε, εργασιακές ενώσεις του προσωπικού, αλλά είναι θέματα τα οποία έχουν επίπτωση στην ε, τεχνική διαχείριση του προσωπικού. Και γι' αυτό το ερώτημά μου προς τον Γενικό Γραμματέα του ελεκτικού συνεδρίου είναι αν υπάρχουν πια πιο αποτελεσματικές διαδικασίες στο ε, ελεκτικό συνέδριο για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις παρενόχλησης του προσωπικού από την διοικητική ιεραρχία. Και αυτό φυσικά συνδέεται με το γενικότερο θέμα του προσωπικού του του ελεκτικού συνεδρίου είχαμε το πρόβλημα ενός θανάτου ενός μέλους του, ενός, ε, μέλους του προσωπικού του ελεκτικού συνεδρίου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδίου στην Πορτογαλία που έλαβε χώρα σε σχέση με μια κοινωνική δραστηριότητα όπως αναφέρεται του ελεκτικού συνεδρίου Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ενισχυθεί η συνεργασία του, συνεργασία του ελεκτικού συνεδρίου με άλλα όργανα. Όταν αυτό οδηγεί στο θάνατο ενός μέλους του προσωπικού, θα ήθελα να ξέρω πώς έγινε κάτι τέτοιο και τι συμπεράσματα μπορείτε να αντλήσετε από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Εάν όχι, Θα ήθελα να έχω τι απαντήσει των ε, θεσμικών οργάνων. Ποιο θα ήθελε να λάβει το λόγο πρώτο στο ελεκτικό συνέδριο, ενδεχομένως. Okay. A few questions for us. Ναι, να απαντήσω στις ερωτήσεις που μας υποβλήθηκαν. Όσον αφορά το κόστος μετάφρασης, εδώ θα το κοιτάξουμε. Πολύ γρήγορα μπορώ να απαντήσω ότι το κόστος ανά σελίδα βασίζεται στο συνολικό κόστος, δηλαδή και ενοικίαση. Το 2012 οι μεταφραστικές υπηρεσίες ήταν σε ένα κτίριο για το οποίο πληρώναμε νίκη, ενώ τώρα έχουν μεταφερθεί στα δικά μας κτίρια. Μπορεί να οφείλεται εκεί η διαφορά. Αλλά θα το κοιτάξουμε και θα σας δώσουμε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, να δούμε κατά πόσο είναι θέμα μεθοδολογίας ή άλλο. Όλα τώρα. Υπάρχει μία περίπτωση που είναι ανοιχτή ακόμα όσον αφορά την Όλαφ. Αλλά εδώ μας καλύπτει το απόρριτο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μόνο που ίσως μπορώ να πω είναι ότι πριν από λίγο καιρό υπήρξε μια επίσκεψη, έκτοτε δεν έχουμε τίποτα νεότερο. Δεν ξέρουμε ποια συνέχεια θα δοθεί. Για περιπτώσεις που εμείς εντοπίσαμε και στείλαμε στην Όλαφ όταν κάνουμε έλεγχο και υποψιαζόμαστε απάτη, σταματάμε τον έλεγχο, ενημερώνουμε την Όλαφ και τότε είναι η Όλαφ η οποία αποφασίζει αν θα ανοίξει ή όχι μια υπόθεση. Το 2005 υπήρξαν 8 περιπτώσεις για τις οποίες ενημερώσαμε την Όλαφ, 6 άνοιξε η Όλαφ και μετά δεν ξέρουμε τι κάνει γιατί Στη στατιστική βέβαια μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις υποθέσεις, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία. Είναι θέματα ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έρχομαι στα μέλη του λεκτικού συνεδρίου και την παρουσία τους στις συνεδριάσεις. Πριν απαντήσω αυτό το συγκεκριμένο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το λεκτικό συνέδριο λειτουργεί με έναν τρόπο που υπάρχουν οι συνεδριάσεις ε, του λεκτικού συνεδρίου αυτού καθεαυτού και μετά των τμήματων συμμετέχουν στα τμήματα, γιατί περισσότερε εκθέσει στα τμήματα εγκρίνονται. Οι μεγάλε συζητήσει δηλαδή ουσιαστικά γίνονται σε επίπεδο τμήματων. Όσον αφορά λοιπόν την παρουσία, κοιτώντα τα νούμερα, κατά τη γνώμη μου δεν δείχνει άσχημη κατάσταση. Γιατί, γιατί τα μέλη κάνουν ε, αποστολές ελεγκτικές, έρχονται εδώ σε εσά. Οπότε η απουσία ενός ή δύο μελών ανασυνεδρίαση από τους 28 είναι κάτι φυσιολογικό. Έρχομαι τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τις διαδικασίες ε, προακογών κλπ. Υπάρχει εναρμόνιση με τα άλλα θεσμικά όργανα γιατί τηρούμε και εμείς τον κανονισμό όλα αυτά, από όσο ξέρω, είναι διαθεσμικά. Δηλαδή έχουμε τους ίδιους εφαρμοστικούς κανόνες. Οπότε αν υπάρχει μια περίπτωση κάποιου που δεν αποδίδει, θα εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό. Όσον αφορά το θάνατο προσωπικού, ναι, υπήρξε μια πολύ ατυχής τέτοια περίπτωση, δυστυχώς. Σχεδόν ήμουν και εγώ σε αυτό το κοινωνικό γεγονός, αλλά πάντως κοινωνική εκδήλωση, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό ήταν το προσωπικό που οργάνωνε την εκδήλωση αυτή. Πριν από τρία χρόνια, για παράδειγμα, πήγα εγώ να παίξω ποδόσφαιρο στην Τσεχία. Δέκα ε, άνθρωποι από το ελεκτικό συνέδριο πήγαν και παίξαν ποδόσφαιρο με άλλες ποδοσφαιρικές ε, ομάδες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ελεκτικό συνέδριο. Υπήρξε έρευνα της αστυνομίας, το αποτέλεσμα πόσο ξέρω δεν κατέδειξε κάποια αδυναμία από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου. Εμείς λίγο πολύ το έχουμε ξεχάσει, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Δεν νομίζω ότι τέθηκε άλλη ερώτηση, αλλά αν θέλετε κάτι παραπάνω, ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψατε τις ερωτήσεις που ήταν για σας. Υπήρχαν ερωτήσεις και για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι. Οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα απαντήσω στις ερωτήσεις που μας ετέθησαν. Καταρχάς, σε σχέση με τη διάρκεια της ε, διαδικασίας ε, και τον ε, αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων. θα ήθελα να πω ότι όλες οι πληροφορίες για το θέμα αυτό υπάρχουν και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ε, που σας αποστήλαμε, όπως και στην ετήσια έκθεση του δικαστηρίου ως οργάνου. Δεν θα ήθελα να δοθεί εντύπωση ότι η διάρκεια της διαδικασίας ε, αυξάνεται ε, σημαντικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν δείτε για παράδειγμα τα προδικαστικά αιτήματα, ερωτήματα που έχουν να κάνουν με εθνικές ε, ε, με εθνικά ζητήματα, κάποια εθνικά δικαστήρια στρέφονται προς το δικαστήριο, το ευρωπαϊκό, για να επιληφθεί του θέματος που τα απασχολεί. Να σας δώσω λοιπόν μία εικόνα. Η, διάρκεια, η μέση διάρκεια της διαδικασίας το 2012 ήταν 15,7 μήνες. Το 2011 ήταν 16,4 μήνες. Το 2009 17,1 το 2007, 19,3. Όσο πηγαίνω προς τα πίσω, η διάρκεια της διαδικασίας αυξάνεται. Οπότε στην πραγματικότητα υπήρξε μείωση της διάρκειας, της μέσης διάρκειας των, ε, της διαδικασίας των προδικαστικών ερωτημάτων ε, κατά την τελευταία περίοδο και το 2012 ισχύει αυτό. Ε, οι άμεσες προσφυγές το 2011 20,2 το 2012 19,7. Ε, θα μπορούσα να σας δώσω μία σειρά αριθμών που δείχνουν ότι η διάρκεια της διαδικασίας ε, μειώνεται παρά το γεγονός ότι σε απόλυτους όρους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αρκετά μεγάλη η διάρκεια αυτή. Υπάρχει και το πρόβλημα της πολυγλωσσίας στο δικαστήριο που επιβραδύνει σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες, ε, γιατί πρέπει να γίνουν μεταφράσεις ε, και αυτό σημαίνει ότι ε, περνάει λίγος χρόνος μέχρι να γίνει και αυτό. Για το ίδιο τώρα το δικαστήριο, ο μέσος όρος τη διαδικασίας, της διάρκειας της διαδικασίας είναι όντως πολύ υψηλός. Είναι πολύ μακρόχρονη διαδικασία. Έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις επί του δικαστηρίου για να γίνει μια προσπάθεια αύξησης παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και να εσπιθευθούν οι διαδικασίες. Ήταν το μέτρο που λάβαμε βέβαια που είχαμε ως ιδέα να λάβουμε ήταν η αύξηση των δικαστών. Γιατί έτσι θα μπορέσει να γίνει η δουλειά μας πιο γρήγορη. Είναι κάτι το οποίο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Εμείς υπολογίζουμε πολύ σε αυτό το μέτρο, Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει και εμείς να λάβουμε κάποια μέτρα από πλευρά μα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας συνεχώς. Για το θέμα της μετάφρασης και της διερμηνίας και το σχετικό κόστος. Η διερμηνία είναι περίπου 80 άτομα. Είναι μάλλον περιορισμένος αριθμός. Οι ακροάσεις μας ε, πρέπει να έχουν διερμηνία λόγω του εσωτερικού κανονισμού. Υπάρχει ένα καθεστώς που διέπει τη διερμηνία, δεν θα μπω σε αλλά μας υποχρεώνει να έχουμε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό διερμηνέων. Όσον αφορά τα χίλια άτομα που δουλεύουν στην πολυγλωσία, εκτός από τα 80 άτομα που ασχολούνται με τη διερμηνία, οι περισσότεροι πάνω από 900 δουλεύουν στη μετάφραση. Ε, σε απόλυτους όρους ε, είναι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων. Να σας εξηγήσω γιατί. Όλη η νομολογία του δικαστηρίου μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες της επίσημης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο είναι ενδεχομένω το μόνο όργανο που ασκεί αυτήν την ε, πολυγλωσία. Και υπάρχει ένας λόγος ότι η νομολογία είναι πηγή δικαίου και η πηγή δικαίου όπως οι συνθήκες, όπως οι κανονισμοί, όπως και οι οδηγίες και επειδή το ε, ουσιαστικό και το παράγωγο δίκαιο ε, είναι ε, πολύ σημαντικά πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες. Πρέπει ο κάθε δικηγόρος να γνωρίζει την ομολογία του δικαστηρίου στη γλώσσα του, ε, είτε είναι Γάλλος είτε είναι ε, Άγγλος. Όλες, ε, όλες, όλα λοιπόν τα συμπεράσματα δημοσιεύονται, κάθε δημοσίευσή μας πρέπει να υπάρχει σε κάθε γλώσσα. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς ε, νομομαθείς ε, νομομαθείς δηλαδή, ε, μεταφραστές. Ε, γιατί πρέπει να μεταφραστούν όλα αυτά σε όλες τις γλώσσες. τα εθνικά δικαστήρια δεν υπόκεινται σε αυτό το περιορισμό της πολυγλωσσίας. Δεν υπάρχουν λοιπόν σε εθνικό επίπεδο υπηρεσίες μετάφρασης, αλλά ήθελα να σας πω ότι αυτή η σύγκριση που μου ζητήσατε να κάνω δεν μου φαίνεται ότι είναι εφικτή. Όσον αφορά την Όλαφ, ναι πράγματι υπάρχει μία έρευνα και θα αναφερθώ σε αυτό. Δεν ε, μπορώ να πω σε ποια φάση βρίσκεται ε, η έρευνα της Όλαφ. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτε ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόστος ε, της μετάφρασης, παρά το γεγονός ότι δεν μας ετέθη το ερώτημα αυτό, είναι αλήθεια ότι όταν είδαμε τα, τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια από τα άλλα όργανα, μας έκανε λίγο εντύπωση ο χαμηλός το, το χαμηλό κόστος το δικό μας σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Και ο λόγος που τον βρήκαμε είναι ότι εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το κόστος του προσωπικού και μόνο. Αν συμπεριβλάβουμε και το έμεσο κόστος, ε, κάναμε βέβαια τότε τους υπολογισμούς, όταν είδαμε τη διαφορά, βρισκόμαστε σε κόστος ανασελίδα 136 ευρώ. Οπότε πλησιάζουμε κατά πολύ το κόστος ε, των υπολείπων οργάνων παρά το γεγονός ε, ότι πρέπει να αναλυθούν ε, λίγο περισσότερο αυτές οι συγκρίσεις γιατί δεν είναι πάντοτε ο ίδιος ο τρόπος εργασίας και όπως είπα και το δικαστήριο έχει νομομαθείς μεταφραστές με μια ιδιαίτερη μέθοδο εργασίας κάτι το οποίο σημαίνει ότι συμμετέχουν πολύ περισσότερο στα ίδια, στην ίδια την παραγωγή ε, εγγράφων από το ε, δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει το κόστος όπως το υπολογίσαμε μετά είναι 136 ευρώ ανασελίδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει τελειώσει η συζήτηση και για το σημείο αυτό. Υπάρχει κάποιο άλλο θεσμικό όργανο που θέλει να λάβει το λόγο. Εάν όχι, Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάμας Δόης, τον συνσηγητή, για την παρουσία του στη συζήτηση. Κλείνει λοιπόν και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους των αλλοθεσμικών οργάνων που ήταν παρόντες σήμερα και έδωσαν τα φώτα τους στη συζήτησή μας. Και μπορώ να κλείσω και αυτό το σημείο της ημέρησης διάταξης. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε σε μία πρωτοβουλία της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και θα κάνουμε σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η, πρωτο, η προθεσμία για τις τροπολογίες τώρα είναι στις την επόμενη εβδομάδα την Τετάρτη. Έχετε μαζί σας το γραπτό κείμενο. Και έχουμε και την ε, θέση του Έλληνα εκπροσώπου του ελεκτικού συνεδρίου. 14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα και η συνάντηση με τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων κρατών, των ελεκτικών αρχών των ε, εμπλεκομένων χωρών. Θα ήθελα να ξέρω τώρα αν κάποιο θέλει να λάβει το λόγο σχετικά. Ο κύριος Γκάιερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία να δω το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε επιφανειακά σε κάποιο επίπεδο. Έχω μονάχα ένα θέμα το οποίο θέλω να εγείρω. Τα σημεία 1 έως 5 υποθέτω ότι μεταφέρουν την προσωπική άποψη του βουλευτού κυρίου Τόιρερ για τα θέματα αυτά, αλλά δεν αποτελούν θέσεις της Επιτροπής μας στο σύνολό της. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι μπορώ να έχω μια διαφορετική θέση για τα θέματα αυτά. σε ό,τι αφορά την ευθύνη των κρατών μελών για την εξέλιξη του χρέους τους. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ευθύνη των κρατών μελών, αλλά της έλλειψη ρύθμισης για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, τουλάχιστον εν μέρη. Αυτά είναι υπεύθυνα για την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό η δική μου προσωπική ομάδα ε, διαφωνεί με τα σημεία 1 έως 5. Φυσικά ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας και γι' αυτό θέλω να προτείνω στον κύριο Τόιρερ να διαγράψει τα σημεία αυτά Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η διαγραφή των πρώτων πέντε σημείων, αλλά έχουμε και προβλήματα με την αντιμετώπιση που έχει γίνει στην Επιτροπή την Οικονομική και Νομισματική και σας λέω αυτό σχεδίως αυτή ήταν, ποια ήταν η πρώτη μου απόψη. Ναι. Προφανώς αυτό θα αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Μα το Κοινοβούλιο δεν έχει να αντιμετωπίσει θέματα της Τρόικα πάντα, γιατί η Τρόικα πολλές φορές αντιμετωπίζει θέματα που ήταν αντικείμενο διμερών συμφωνιών και συμφωνών με την ε, Κεντρική Τράπεζα, των Εθνικών Τραπεζών με την Κεντρική Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά κάνει μια τεράστια επίθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μπορεί να εξυπηρετήσει τους προεκλογικούς στόχους ορισμένων. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το θετικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα περιττή μια τέτοια γνωμοδότηση από τη δική μου, από τη δική μας Επιτροπή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να διακριβώσουμε γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν απορροφήσει τα κονδύλια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την κρίση. Το θέμα της αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης σε 90% δεν έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη απορρόφηση. Γιατί λοιπόν παραμένει προβληματική αυτή η απορρόφηση, αυτή η διαρθρωτική αλλαγή. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας αντιμετωπίσει. Γιατί η Κομισιόν έχει επιτρέψει μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι μέλος κράτος 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο έχει νόημα για μένα. Όλη αυτή η έκθεση για την Τρόπικα Τρόικα νομίζω ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτά που είναι εδώ πέρα διατυπωμένα στην έκθεση αυτή για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο αυτό δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να τα υποστηρίξω. Δεν είναι θέμα βελτίωσης και καλοπισμού της διατύπωσης. Νομίζω ότι όπως και πολλά άλλα στοιχεία της εργασίας μας δεν ε, αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα σοβαρότητα. δεν πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στις χώρες κρίσης ότι αρκετά έχετε κάνει και δεν πρέπει να κάνετε περαιτέρω προσπάθειες. Αυτό είναι ένα λανθασμένο μήνυμα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα και γι' αυτό εγώ δεν μπορώ παρά να πω ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπαθίε τους και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα με τη δική μας ε, Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ προβληματικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παραγνωρίσει κανείς τις προσπάθειες χωρών όπως η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να επιρρύψει την ευθύνη σε χώρες όπως η Γερμανία. Επομένως, νομίζω ότι ήδη η πρώτη παράγραφος έχει νόημα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες διατυπώσεις, γιατί έχουμε μία γνωμοδότηση εμείς θα έπρεπε να επικεντρωθούμε μονάχα στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να καταθέσει τροπολογίες για να περιορίσει την γνωμοδότηση στα θέματα της Επιτροπής, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην υπάρξει καν και μια γνωμοδότηση από τη δική μας πλευρά. Αυτά. Ευχαριστώ. Έχουμε ως Επιτροπή μερικές φορές την εντύπωση ότι ορισμένες φορές δραματοποιούνται ορισμένα θέματα. Το θέμα της Τρόικας είναι ένα συγκεκριμένο και σημαντικό θέμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε απαραίτητη η δράση της ε, Τρόικα για ορισμένα κράτη-μέλη. Δεν μπορούσε κανείς να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να δεχτούν την Τρόικα. Το έκαναν με δική τους απόφαση. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να δοθούν οι απαραίτητες εγγύησεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και αυτές οι βοήθειες που δόθηκαν συνδεόταν με το ρόλο της Τρόικα. Μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα του αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει μια άποψη για τα θέματα αυτά. Αλλά είμαστε ε, ένα ελεύθερα εκλεγμένο ε, όργανο και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Έγινε μια ακρόαση για το θέμα της ε, Ελλάδος. Ε, πρόκειται να γίνει μάλλον το, μια ακρόαση η οποία αναβλήθηκε με προ, πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της ε, Task Force της Κομισιόν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες κρίσης. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ καταλαβαίνω, το λέω από την αρχή, ότι αυτή η γνωμοδότηση έχει προκύψει κάτω από μεγάλη χρονική πίεση και Δυστυχώς μέχρι την, ε, τα Χριστούγεννα δεν είχαμε ακόμα το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να μπορέσουμε να καθορίσουμε καλύτερα την εργασία μας. Αλλά κύριε Γκάιερ, ιδίω στο σημείο 1 και στο σημείο 5 αυτά τα οποία αναφέρονται είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο προέκυψε από τη διακοινοβουλευτική συνάντηση και από τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικα, γιατί στην διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ετέθη πράγματι το θέμα του κατά πόσο οι ελεκτικές ικανότητες του κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου είναι επαρκείς για να μπορέσουν να αποτρέψουν μια τέτοια κρίση όπως αυτή που αντιμετωπίζουν ορισμένε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει ένα συνολικό δημόσιο χρέος 175% του ΑΕΠ, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει προκληθεί το χρέος αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το Εθνικό Κοινοβούλιο που δέχτηκε τα απαραίτητα μέτρα που οδήγησαν σε αυτό το μεγάλο χρέος. Θα μπορούσε να είχε πει το Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα τόσο μεγάλο χρέος και θα μπορούσε με τις αποφάσεις του το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ε, απορρίψει αυτή την υπερβολική υποχρέωση. Υπάρχει αυτό το ερώτημα λοιπόν που έχει να κάνει με το παρελθόν. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον και να τι αποτρέψουμε. Το θέμα του ελέγχου του προπολογισμού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι η δική μα αρμοδιότητα και είναι σημαντικό όταν γίνεται αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε τις επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν για τις συγκεκριμένες δαπάνε. και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της οικονομικής συγκυρίας. Η δική μας επιτροπή είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια για να πει με ποιο τρόπο θα γίνεται η καλύτερη ε, λειτουργία του δημοσιονομικού ελέγχου και η καλύτερη χρησιμοποίηση των χρημάτων. Εμείς είχαμε και την αρμοδιότητα και την εμπειρογνωμοσύνη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Αν εμείς οι ίδιοι που είμαστε στην καλύτερη θέση λοιπόν να ασκήσουμε το δημοσιονομικό έλεγχο αποσύσουμε την ευθύνη να αναφερθούμε για τα θέματα αυτά, εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία αυτή η οποία ανοίγεται για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε τις σωστές θέσεις για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει ο έλεγχος από την επερχόμενη Επιτροπή του Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δώσουμε μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων όπως έχουμε υποσχεθεί και φυσικά εγώ μπορώ να αποδεχθώ <laughs> ότι η διατύπωση αυτού του κειμένου σίγουρα έχει οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις. Ο Σέρεν. Ευχαριστώ. Δεν είχα φανταστεί στην αρχή ότι θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα μπω τελικά. Αυτά που λέει το Κοινοβούλιο όμως δεν νομίζω ότι είναι σωστά. Μπορούμε να κάνουμε μια δήλωση ξεκινώντα από την Ελλάδα, αλλά θα ήταν πιο σωστό να ξέρουμε ότι όλες οι χώρες πλήττονται από τη δημοσιονομική κρίση. Μια χώρα σαν την Ιρλανδία ή μια χώρα όπως η Ισπανία δεν πλήττονται. Το γεγονός ότι τηρούν όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πού οδήγησε τελικά το έλλειμμα αυτό δημιουργήθηκε επειδή έπρεπε να σώσουν τις τράπεζες. Και γιατί έπρεπε να σώσουν τις τράπεζες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτησε, γιατί φοβήθηκε ότι η κρίση αυτή στην Ιρλανδία η τραπεζική θα διαδόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε δεν είναι σωστά αυτά που λέγονται εδώ. Μπορούμε γενικά να γράψουμε μια έκθεση για την Ελλάδα και να πάρουμε σημείο κίνηση στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι σωστό όταν σκεφτούμε την Ισπανία ή την Ιρλανδία. Εκεί ήταν περισσότερο θέμα ελέγχου τραπεζών και όχι ελέγχου των ε, δημοσιονομικών των χωρών. Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης τώρα. Äh, Έχει δίκιο σε ένα σημείο ο Σόρεν. Σίγουρα το παράδειγμα της Ιρλανδίας καταδεικνύει ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο των τραπεζών, όπως είπε ο Σόρεν. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ένα είδος φυσικής καταστροφής που ενέσκυψε πάνω στις ε, χώρες αυτές και για την περίπτωση της Ελλάδος δεν είναι σωστό ότι η Ελλάδα ήταν απόλυτα υπεύθυνη για το χρέος της. Άμα δει πόσο βομβαρδίστηκαν οι Έλληνες πολίτες με ευνοϊκές προτάσεις από τις τράπεζες με χαμηλά επιτόκια για το δεύτερο αυτοκίνητο, το τρίτο σπίτι κτλ. Υπήρξε μια τεράστια πίεση που ασκήθηκε από την πολιτική χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ουσιαστικά οδήγησε τα κεφάλαια με πολύ φθηνά επιτόκια στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Υπήρξε λοιπόν μια πίεση από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια Ευρώπη για μεταφορά κεφαλαίων σε χαμηλά επιτόκια που έπαιξε και αυτή κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό. Όταν όμως εμείς περι αντιμετωπίσουμε το θέμα του ελέγχου του προπολογισμού θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι προϋπολογισμοί και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού σε ορισμένες χώρες είναι κάτι το οποίο δεν θα μας ενδιαφέρει και το λέω σαφώς. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας απαντώντας σε μια ερώτηση του κυρίου Πόστ τον Ιούλιο του 2013 και η απάντηση δόθηκε πριν από τις εκλογές είπε ο Βολφγαν Σόιμπλε ως Υπουργό Οικονομικών ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας έχει λόγω των χαμηλών επιτοκίων στην Γερμανία και των υψηλών επιτοκίων στην Ισπανία, την Ιταλία και άλλων χωρών, είχε εξοικονόμηση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα μεγάλο ποσό. Ενώ το ποσό το οποίο έχει δοθεί από τη Γερμανία για τη, διάσωση άλλων χωρών δεν ξεπερνάει τα 35-40 δισεκατομμύρια. Η Γερμανία έχει εξοικονομήσει λοιπόν 140 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι χρήματα τα οποία πρέπει να θεωρηθούν καθαρό κέρδος της Γερμανίας. Εάν δεν είχε υπάρξει η κρίση στην ε, Ευρωζώνη, αν δεν υπήρχε η αρνητική αντιμετώπιση από τις αγορές τη της Γερμανίας και της Ισπανίας, θα είχε μαζέψει λοιπόν η Γερμανία αυτά τα κέρδη. Μήπως πρέπει αυτά τα γερμανικά κέρδη να θεωρηθούν ευρωπαϊκά κέρδη. Γι' αυτό ε, νομίζω ότι η δυσκολία με το σημείο 1 είναι ότι δεν περιλαμβάνει καθόλου τέτοιου είδους στοιχεία. Ξέρω ότι πηγαίνει ο Φρανκ Βάλτερ Μάρες στην Αθήνα σήμερα για να συζητήσει ακριβώς για αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να υπάρχει υπερκέρδος για ορισμένα κράτη και φυσικά είναι δύσκολο να αναδιανεμηθούν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση για να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση των χωρών κρίσεων. Γι' αυτό είναι απαραίτητο στην παράγραφο αυτό να τονίσουμε για την ε, συνολική ευθύνη η οποία υπήρξε και το γεγονός ότι ορισμένες χώρες επωφελήθηκαν από αυτή την κρίση. Και επίσης επανέρχομαι στο σημείο αυτό που αναφέρει ότι η Τρόικα είναι ένα τεχνοκρατικό σώμα, γιατί η Τρόικα η θελημένα δεν έχει παίξει καθαρά τεχνοκρατικό ρόλο αλλά έχει παίξει ένα ρόλο που θα τον χαρακτήριζα ως πολιτικο-ιδεολογικό σε ορισμένε περιπτώσεις. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα να ακολουθούμε μια λαθασμένη πολιτική. Το πρώτο με μνημόνιο για την Ελλάδα ήταν απόλυτα λανθασμένο, βασιζόταν σε λαθασμένες παραμέτρους και συνεχίζεται παρόλα αυτά η δραστή στρόικα. Αυτό για ιδεολογικούς λόγους. Επομένως πρέπει να βγάλουμε την έκφραση τεχνοκρατικό ή τεχνικό σώμα και νομίζω ότι το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης δεν ήταν απλώς ένα ασθενές σημείο. Ήταν απόλυτα απούσα η δημοκρατική νομιμοποίηση. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να έχουμε εγκαίρως μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει την ε, Τρόικα. Σήμερα ο ο Ότμαρ Κάρα και ο Γάλλο συνάδελφό σα από του σοσιαλιστέ θα πήγαιναν, θα έπρεπε να πάνε στην Αθήνα. Δεν πήγαν τελικά. Έχει αναβληθεί αυτό το ταξίδι. Η ΕΚΟΝ Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια υποεπιτροπή για να αντιμετωπίσει το θέμα τη Τρόικα. Αλλά θα έρθει αυτό το, η έκθεσή τη πολύ αργά πια τον Απρίλιο όταν θα φεύγει το Κοινοβούλιο, θα πάει να λειτουργεί. Επομένως υπήρξε μια έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης για την ε, ε, Τρόικα και το τελευταίο, τελευταία παράγωση που λέει ότι χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι μια οραματιστική προσέγγιση που πρέπει να την υποστηρίξουμε. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Εγώ χαίρομαι να, που κατάφερα να προκαλέσω με αυτό το έγγραφο μια πολιτική συζήτηση στην Επιτροπή. Είναι μια πολιτική συζήτηση, λέει ο κύριος Γκάιερ, Εγώ νομίζω ότι η ουσία σε αυτά τα θέματα είναι μια υπόθεση της Οικονομικής Επιτροπής και εδώ βρίσκεται και η τυπική μου αντίρρηση. Ο Σόρεν είπε πολλά πράγματα που ήθελα να πω και εγώ. Και για τον Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεσαι τώρα στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα και θα είσαι μαζί μας στα θέματα αυτά. Τουλάχιστον σε αυτό το θέμα υπάρχει μια πολιτική συμφωνία. Πάντως παραμένει το θέμα του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε πολιτικό επίπεδο την Τρόικα. Βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να πει κάτι για το θέμα αυτό γιατί είμαστε ένας πολιτικός οργανισμός. Και αυτός είναι και ένας χώρος ο οποίος είναι πολιτικού χαρακτήρα και εμπλέκει και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα έπρεπε να έχει και μια αρμόδια ε, ένα αρμόδιο όργανο το οποίο να λάβει θέση για τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το έγγραφο, την πρόταση γνωμοδότησης του Μίχελ Τόιερ που πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι για το οποίο επικρίνουμε άλλες ε, επιτροπές. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για την πολιτική αντιπαράθεση Είμαστε μια επιτροπή η οποία έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για τα θέματα αυτά, μπορεί να την εκφράσει στην Ολομέλεια σε άλλους χώρους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τα τεχνικά θέματα της Επιτροπής μας από τις πολιτικές θέσεις και να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία είναι τα δικά μας θέματα και παραμένω σε αυτό το σημείο ότι πολλά από τα κομμάτια της ε, γνωμοδότησης αυτής, του σχεδίου γνωμοδότησης, δεν έχουν καμία σχέση με τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει τη διαγραφή τους. Σε αυτά που είπες για την ε, διάσκεψη με τα εθνικά κοινοβούλια. Βεβαίως. Μπορούμε θαυμάσια να το αναφέρουμε αυτό ότι έγινε αυτή η συνδιάσκεψη και λαμβάνουμε υπόψη τα συμπεράσματα αυτής της ε, συνδιάσκεψης. Αυτό μπορεί να κάνει σαφές και γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε κάποια γνωμοδότηση και είμαι έτοιμο να σε βοηθήσω να βρει μια διατύπωση η οποία θα καλύπτει αυτά τα σημεία. Ο Γιάννη Μιλντόρ. Το θέμα είναι τόσο περίπλοκο που μέχρι τώρα σώπασα. Άκουσα μόνο τα επιχειρήματα. Όμως, αν δούμε το σημείο 1, το κύριο πρόβλημα είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία δεν φτιάχτηκε βάσει μιας καθορισμένης κοινωτικής μεθόδου. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να αυτολέγχονται. Και αυτή είναι η κύρια αιτία του προβλήματος. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Από τη στιγμή που διαπραγματευόμαστε για μια τραπεζική ένωση, το ίδιο πρόβλημα επανέρχεται συνεχώς. Διαδικασία απόφασης. Και αυτό είναι νομίζω το πρόβλημα που πρέπει να ελέγξουμε και εδώ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα που να συνάδει με τις καθιερωμένες διαδικασίες, γιατί η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ανεξαρτησία. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αναμειχθεί. Είναι βασικός ο ρόλος της, στην επίλυση της κρίσης, οπότε ειλικρινά δεν μπορώ να βρω την σωστή διατύπωση, αλλά για πείτε μου ποια είναι η πρόθεσή σας. Νομίζετε ότι μπορούμε να το τροποποιήσουμε αυτό το κείμενο, τι σκοπεύετε να κάνετε. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, ε, σας παρακαλώ όλους να υποβάλλετε τροπολογίες. Η συζήτηση που κάναμε εδώ έδειξε ότι υπάρχουν κοινέ απόψεις, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, πολιτικές διαφωνίες. Μια που είχαμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε, παραδέχομαι κι εγώ ότι υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις εδώ που ήξερα ότι θα προκαλούσαν τη συζήτηση. Συνεπώς, ποια είναι η πρόθεσή μου. Η πρόθεσή μου είναι το εξή. Είμαι πεπισμένο ότι η άποψη τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών πρέπει να συμπεριληφθεί στην ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων ή στη συζήτηση για αλλαγή του κανονισμού όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κρίση, τότε διαπιστώνουμε ότι η δημοσιονομική κρίση στις χώρες μέλη δεν έχει Έχει επιπτώσεις τελικά υπάρχουν επιπτώσεις στην, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό προφανώς για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν τα κονδύλια. Άρα είναι θέμα ελέγχου προπολογισμού. Και υπάρχουν και επιπτώσεις στον EFSM από τον κοινοτικό προπολογισμό. Οπότε το ζήτημα είναι ποιος τελικά ελέγχει τον μηχανισμό αυτόν, ποιος τον εποπτεύει. Αν λοιπόν το δείτε καλά, υπάρχουν πτυχέ ελέγχου προπολογισμού. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι περισσότεροι θέλουν να μα κρατήσουν εκτό. Και ακόμα και με αυτόν τον μηχανισμό default που αναρωτιόμουν κατά πόσο έπρεπε ή όχι να το συμπεριλάβουμε και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί τα εθνικά δημοσιονομικά θεωρούνται υπεύθυνα για την κρίση γιατί δεν είναι ένας ε, τέτοιος μηχανισμός default. Οπότε γι' αυτό πιστεύω και εγώ ότι είναι θέμα ελέγχου προπολογισμού. Πώς θα αποφύγουμε τις επιπτώσεις στο κοινοτικό προπολογισμό μόνο αν καταφέρουμε να αναπτύξουμε παρετέρω έναν μηχανισμό των ε, χωρών όπου να συμμετέχουν οι ιδιωτικοί δανειστές, να αναλαμβάνουν και αυτοί δηλαδή το κίνδυνο και να συμμετέχουν στη λύση στην περίπτωση κρίσης. Νομίζω λοιπόν για όλα αυτά τα σημεία στη γνωμοδότηση μπορεί να μην ε, μας βρουν σύμφωνους, αλλά ας περιπτώσει θα συνεχιστεί η συζήτηση. Προτείνω λοιπόν να έχω μια συνάντηση με τους σκιώδες εισηγητές στο Στρασβούργο ίσως. Αν συμφωνείτε ή αλλιώς αν μου στείλετε τροπολογίες, μια διαφορετική διατύπωση, θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη μου ό,τι προτείνατε που έχουν να κάνουν με το θέμα διακοινοβουλευτικά θα προσπαθήσω να τα προωθήσω και να αποδείξω έτσι στο Κοινοβούλιο ότι η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με την Επιτροπή μας. Καλώς. Ωραία. Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Συμπεραίνω πως Ολοκληρώνεται προς το παρόν η συζήτηση για αυτό το θέμα, αν δεν έχει κανείς άλλος τίποτα να προσθέσει. Η προθεσμία. Την Τετάρτη 15 του μηνός είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. the point of this approval of the uh, mm. to the joint uh, yep. statement okay. from the three institutions mm -hmm. that we put yep. in coordinators at the last okay. moment yesterday. Ich schließe damit die Επομένως μπορώ να κλείσω την συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ελέγχου του προϋπολογισμού. Απλώς πρέπει οι συντονιστές να κάνουν μια εξέταση ορισμένων σημείων πριν από τη δεξίωση την οποία σας έχω προσκαλέσει μαζί με τους συνεργάτες μας και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συντονιστές να παραμείνουν εδώ για να κάνουμε την συνεδρία των συντονιστών.